στην Ολομέλεια. Είναι η πρώτη σας ομιλία, κυρία Πρόεδρε, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε συμφωνήσαμε να σας δώσουμε περισσότερο χρόνο, γιατί ο κύριος Πρόεδρος θέλει να σας εκθέσει τις απόψεις του και για άλλα θέματα και θεσμικά κατά την έναρξη της θητείας του. Οπότε ελπίζω να αρκεστείτε σε 15 με 20 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχω αυτή τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε μια συζήτηση μαζί σας. Όχι μόνο να αναφερθώ στην ανεπίσημη συνοδοκορυφή που έγινε από δύο εβδομάδες. Ήταν ανεπίσημη συνάντηση εξάλλου. Δεν υπάρχουν επίσημα συμπεράσματα αλλά δράτω με τις ευκαιρίες για να συναντηθώ μαζί σας στις αρχές της θητείας μου. Αν περίμενα μέχρι την πρώτη επίσημη δυνατότητα να αναφερθώ στα όσα γίνονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τέλος Μαρτίου, δεν θα ερχόμουν στο Κοινοβούλιο πριν από το τέλος Απριλίου. Πέντε μήνες λοιπόν μετά το διορισμό μου στη θέση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν να περιγράψω το ρόλο μου, τα καθήκοντά μου, πώς τα βλέπω εγώ. Θα μιλήσω για λίγα λεπτά πάνω σε αυτό. Για να μην επιστρέψω αυτά τα θέματα σε μελλοντικέ ευκαιρίε. Πάντα υπήρχε Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν είναι το ίδιο με τον Πρόεδρο του, της Ευρώπης όπως αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης. Τι άλλαξε. Τρία μικρά πράγματα τα οποία με την παρόδο του χρόνου όμως όλα μαζί θα οδηγήσουν στη μεγάλη διαφορά. Πρώτα απ' όλα έχουμε το στοιχείο της συνέχειας. Η, κατά το παρελθόν άλλαζε κάθε εξάμενο η Προεδρία. Κάθε δεύτερη τρίτη συνεδρίαση του Συμβουλίου λοιπόν. Άρα δεν υπήρχε δυνατότητα για διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Οι εταίροι μας σε τρίτες χώρες προβληματιζόταν διότι συναντούσαν διαφορετικό αρχηγό κυβερνήσεως κάθε φορά που διεξαγόταν μια σύνοδος κορυφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνέχεια είναι θεμελιώδου σημασίας για την οικοδόμηση σχέσεων και για την επίτευξη σοβαρών καθηκόντων και στόχων. Δεύτερον, αυτή η πλήρης απασχόλησης είναι διαφορετική. Προηγούμενοι πρόεδροι έπρεπε να χειρίζονται και την εθνική τους κυβέρνηση ταυτόχρονα αυτό το καθήκον θα μπορούσαν να το μοιράζονται μόνο με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, να μοιράζονται το χρόνο τους. Δημιουργώντας μια θέση αποκλειστική που αφορά το, τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση Ευρώπης προς τα έξω, με αυτό το ρόλο μπορεί να παίξει καλύτερο ρόλο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εντός του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Συστήματος. Τρίτον, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιλέγουν ποιος θέλουν να κατέχει αυτή τη θέση. Να μην συμβαίνει τυχαία μέσω ενός αυθαίρετου ε, συστήματος εναλλαγής. Πιστεύω ότι αυτός είναι καλός ιονός για την υποστήριξη που ελπίζω να τύχει ο Πρόεδρος. Αυτές οι τρεις αλλαγές είναι πραγματιστικές βελτιώσεις όσον αφορά την πρώτερη θεσμική αρχιτεκτονική. Όλα αυτά μαζί με το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γίνεται θεσμικό όργανο Αυτά δίνουν καλύτερες δυνατότητες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εκπληρώσει τους στόχους του, που απορρέουν από τις συνθήκες που καθορίζουν τις γενικές, γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Ενώσεως. Κάποιοι σχολιαστές είδαν ότι περιέχει πολλά περισσότερα αυτός ο ρόλος. Κάποιοι είδαν ότι περιέχει λιγότερα. Από τη μία πλευρά, κάποιοι θεωρούν την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σαν ένα είδος προέδρου. Δηλαδή, με εκτελεστική εξουσία επικεφαλής ενός κράτους όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας. Άλλοι βλέπουν αυτή τη θέση σαν απλή θέση Προέδρου του Συμβουλίου των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Στην πραγματικότητα δεν είναι κανένα από τα δύο. Σίγουρα δεν είναι πρεζιντό, δεν είναι Πρόεδρος που έχει εκτελεστικές εξουσίες από μόνος του. Θα πρέπει ο κάτοχος της θέσης να εκφράζει τις απόψεις όλων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Από την άλλη πλευρά ο ρόλος του δεν είναι απλώς ο ρόλος ενός Προέδρου που δίνει το λόγο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να μιλήσουν κατά τη διάρκεια των συνόδων αυτών. Χρειάζεται να προετοιμάζει τις συνεδριάσεις, να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις και να εκπροσωπεί την Ένωση στο εξωτερικό μαζί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη Συνόδου του G20 και είναι γέφυρα μεταξύ εθνικών πρωτευουσών και θεσμικών οργάνων όλα αυτά ξεπερνούν σαφώς το καθήκον ε, απλού Προέδρου μιας συνεδρίασης. Ο ρόλος του μονίμου Προέδρου είναι να δίνει ένα ισχυρό συνέστημα κατεύθυνσης. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Πού πηγαίνουμε, πώς αντιμετωπίζουμε τους γειτονές μας, ποια είναι η βασική μας στρατηγική εταίρη στον κόσμο, πού θέλουμε να είμαστε σε 10-20 χρόνια. Αυτά είναι ζωτικά θέματα. Όσον αφορά τη σχέση μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συνθήκη είναι αρκετά σύντομη όσον αφορά το θέμα αυτό. Απαιτεί απλώ να έρχομαι και να σα ενημερώνω μετά από συνεδριάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ένα ελάχιστο τέσσερι φορέ το χρόνο. Τα περισσότερα χρόνια πιθανότατα θα είναι πέντε, έξι φορέ και ίσω να φτάσουμε και στι δέκα φορέ το χρόνο. Σύντομα, πολλοί από εσά θα βαρεθείτε να με βλέπετε. Θα συνεχίσω να πολλαπλασιάζω τις επαφές μου με τα μέλη του Κοινοβουλίου με συναντήσεις προέδρων ομάδων και μηνύα συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ρόλος μου πράγματι δεν θα πρέπει να συγχέεται με το ρόλο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Μπαρόσο ηγείται εκτελεστικού κλάδου που εκλέγεται και είναι υπόλογο το σώμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλει νομοθετικέ και δημοσιονομικέ προτάσει, προτάσει του προπολογισμού. Εγώ δεν κάνω κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθημερινή επαφή, στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεργάζεται μάλιστα επί θεμάτων νομοθετικού περιεχομένου και όσον αφορά τον προπολογισμό. Το καθήκον μου είναι να εξασφαλίζω ότι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μπορούν συλλογικά να συμφωνούν επί γενική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά την εσωτερική ανάπτυξη αυτής και όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις αυτής. Σε εβδομαδία συνάντηση με τον κύριο Μπαρόσο γνωρίζουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση καθηκόντων μεταξύ μας και παρεξηγήσεις ποιο είναι υπεύθυνο γιατί. Η κοινή γνώμη και οι τρίτες χώρες θα έχουν δυσκολίες να δουν ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχω πεποίθηση όμως ότι ακολουθούμε το σωστό δρόμο για να μην συμβεί αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να θυμηθούμε κάτι ότι είμαι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όχι του Συμβουλίου Υπουργών. Αυτά είναι ξεχωριστά θεσμικά όργανα. Το κανονικό Συμβούλιο που είναι ο άλλος κλάδος ο νομοθετικός μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξακολουθεί να προεδρεύεται από μια προεδρία που θα εξακολουθεί να εναλλάσσεται ανά ε, και να αναλαμβάνει κάθε φορά ένα κράτος μέλος μόνο στη μορφή του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου συντονίζεται η εκτελεστική εξουσία, υπάρχει μόνιμος πρόεδρος υπό τη μορφή της Κάθριν Άστον, που είναι αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι εκπρόσωπος για εξωτερική πολιτική της Ενώσεω. Θα σταθώ εδώ για να αποτίσω φόρο τιμής στη δουλειά που έκανε η Κάθριν Άστον. αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας και προετοιμάζει την εξωτερική δράση, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και πρέπει να τη στηρίξουμε. Θα είναι προνόμιό μου να συνεργαστώ στενά μαζί της όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση της Ενώσεως. Να πω μερικά λόγια για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το ίδιο. Η πρώτη επίσημη συνεδρίαση υπό την Προεδρία μου θα λάβει χώρα τέλος του επομένου μηνός όμως έγινε μια σύνοδος ανεπίσημη αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων αρχές του έτους στην βιβλιοθήκη Σολβέ, μερικές εκατοντάδες μέτρα από εδώ. Τώρα, λόγω του κλίματος της βιβλιοθήκης ή επειδή ήταν κοντά το κοινοβούλιο δεν ξέρω αλλά ήταν καρποφόρες οι συζητήσεις μας όπως είπα δεν μπορώ να σας ενημερώσω όσον αφορά επίσημα συμπεράσματα διότι ήταν ανεπίσημη αυτή η σύνοδος το πολύ μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τις δικές μου προσωπικές απόψεις και τα συμπεράσματά μου από τις συζητήσεις. Τα συμπεριέλαβα αυτά σε μια επιστολή που έστειλα προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το γράμμα αυτό έχει διανεμηθεί και, στην, στο Κοινοβούλιο. Στόχος μου με το ανεπίσημο αυτό συμβούλιο ποιος ήταν να προετοιμάσω τις μελλοντικέ μας συζητήσεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις οικονομικές επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσων εξερχόμεθα από την οικονομική κρίση. Άρα πρέπει να δούμε ποια θα είναι οι στόχοι μας, ποιες θα είναι οι φιλοδοξίες μας. Και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μπαρόσο, μας έδωσε ένα χρησιμότο έγγραφο πάνω σε αυτό. Και επίσης θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διακυβέρνησή μας όσον αφορά αυτά τα θέματα. Πώς μπορούμε να χειριστούμε την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή οικονομία που είναι η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Ούτως ώστε να βελτιώσουμε τις οικονομικές μας επιδόσεις που είναι ένα από τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχική ανταλλαγή απόψεων επ' αυτών συνεπάγεται την εξέταση του καθορισμού στόχων, πώς επιτυγάνονται οι στόχοι και πώς αξιολογούνται τα αποτελέσματα. Κατά πολύ αυτό αφορά το συντονισμό των προσπαθειών που ασκούν τα κράτη-μέλη, χρησιμοποιώντας πλήρως και τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωση και τα διάφορα συναφή μέσα. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι πολύ ταιριαστό για να τα κάνει όλα αυτά. Στη συνεδρίαση του Σολβέ, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμφώνησαν ότι χρειαζόμαστε καλύτερη, πιο εστιασμένη οικονομική προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο συντονισμένη και μακροοικονομικά, για μακροοικονομική πολιτική στην Ευρωζώνη και για μικροοικονομική πολιτική. Πολλά από αυτά είναι πολύ τεχνικής φύσεως, αλλά ας δούμε ποια είναι η ιδέα να μειωθεί ο αριθμός των κοινών οικονομικών στόχων και να επικεντρωθούμε επί τεσσάρων ή πέντε τέτοιων στόχων. Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να είναι ποσοτικοποιημένοι και ορατοί σε εθνικούς υποστόχους. Δεν έχει νόημα να έχουμε βαθμολόγηση 65 ξεχωριστών στόχων. Και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θέλουν να υπομισθούν περισσότερε ευθύνε όσον αφορά μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Τέτοια προσωπική εμπλοκή και προσπάθεια είναι απαραίτητη. Πρέπει από επι επιχάρτου να πάμε σε πραγματικέ, ρεαλιστικέ δεσμεύσει Και χάρηκα που είδα ότι υπάρχουν τι φιλοδοξίε γύρω το τραπέζι. Τώρα, να το αποκαλέσουμε καλύτερο συντονισμό, καλύτερη διακυβέρνηση ή gouvernement économique. Βασικό είναι να θέλουμε όλοι να πετύχουμε. Επίσης, συζητήσαμε εντάχει πώς να εφαρμόσουμε καλύτερα τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την ανοικοδόμηση της ΑΙΤΙΣ. Θέλουμε να προχωρήσουν συζητήσεις ούτως ώστε να εφαρμόσουμε καλύτερα το άρθρο 214 της Συνθήκης όσον αφορά το συντονισμό στην ανθρωπιστική βοήθεια μια συζήτηση για το πώς η Ευρώπη θα μπορούσε να δώσει στατικές απαντήσεις στη διάσκεψη της Κοπενχάγης για την αλλαγή του κλίματος θα είναι κάτι που θα συζητηθεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Απροσδόκητα βέβαια έγινε και συζήτηση για την κατάσταση στην Ελλάδα και εγώ ανέλαβα ο ίδιος προσωπικά να διαβεβαιώσω ότι θα εξεταστούν όλα αυτά στο θεσμικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στα ζητήματα τη Ελλάδο και όχι εκτό του θεσμικού πλαισίου. Και ότι η συμφωνία που επετεύχθη με την έγκριση και των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, καθώ και με τη συμφωνία του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτή η συνένεση ήταν ένα μήνυμα για την αποδοχή από πλευρά Ελλάδα των ευθυνών για να περικόψει κατά αξιόπιστο τρόπο την, το έλλειμμά τη και την αλληλεγγύη που δείχνουμε έναντι τη Ελλάδο αν χρειαστεί. Προσβλέπω στο να ακούσω τι απόψει σα επί όλων αυτών των ζητημάτων και μάλιστα κατά πόσο, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που ε, περιμένουν την Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας διαβεβαιώνω ότι έχω έναν βασικό στόχο για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να εξασφαλίσω το ότι η Ένωσή μας θα είναι αρκετά ισχυρή εσωτερικά. Θα διατηρήσει το δικό μας κοινωνικό μοντέλο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό θα προσπιστούμε τα συμφέροντά μας και θα προβάλλουμε τις αξίες μας. Νομίζω ότι όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν και θα πρέπει να συνεργαστούν για την επίτευξη αυτών των στόχων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Τώρα θα ακούσουμε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχάς να συγχαρώ τον Πρόεδρο Βαν Ρομπόη για την πολύ καλή ανεπίσημη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έγινε για πρώτη φορά υπό την Προεδρία του. Αφού καταλήξαμε στη συμφωνία όσον αφορά τη σημαντική δήλωση για την Ελλάδα, συζητήσαμε τη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020, στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Είχα τη δυνατότητα, έχω τη δυνατότητα να εστιαστώ επί ουσιαστικών θεμάτων που αντιμετωπίζουμε στην πολιτική μας, σε σχέση με αυτές τις προκλήσεις και θα υποβάλουμε κάποια θέματα την επόμενη Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημα. Πριν από την κρίση, η ευρωπαϊκή οικονομία πρόδευε. 18 εκατομμύρια νέε θέσει απασχόληση, πιο δυναμικό περιβάλλον επιχειρηματικό δημιουργήθηκε, αλλά αυτά τα κέρδη τελικά εξαλείφθησαν από την χρηματοπιστωτική κρίση και από τι συνέπειε που είχε σε πολλού τομεί δραστηριοτήτων. 4% μείωση του ΑΕΠ σε ένα χρόνο, ανεργία που έφτασε το 10%, τεράστιο πλήγμα προς την ευμάρειά μας, πραγματική απειλή για τις κοινωνίες μας. Ταυτόχρονα ο στόχος γίνεται δυσκολότερος. Έχουμε κοντά πληθυσμό, αυξανόμενη διαφορά παραγωγικότητας με τους ανταγωνιστές μας και διάφορα κενά όσον αφορά την έρευνα και την παιδεία. Έχουμε όμως και ισχυρά σημεία. Έχουμε τη μεγαλύτερη οικονομία της αγοράς του κόσμου, έχουμε την ενιαία αγορά, έχουμε την Ευρωζώνη, και όλα αυτά απεδείχθησαν σημαντικό στοιχείο ενεργητικού στην κρίση. Αλλά σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολύ σημαντική επιλογή, θα έλεγα σχεδόν καθοριστική επιλογή για το μέλλον των νέων γενεών. Ελπίζοντας για μια επιστροφή στις παλιές καλές μέρες, αυτό δεν είναι μια επιλογή, δεν θα επιστρέψουν. Μια επιλογή είναι περιορισμένες αλλαγές ο ελάχιστο κοινό παρονομαστή που επιφέρει κάποια ανάπτυξη, κάποιε μεταρρυθμίσει, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε αυτά που χάσαμε στην κρίση. Αυτή η επιλογή θα οδηγούσε σε μια Ευρώπη που θα είναι στη δεύτερη κατηγορία τη νέα παγκόσμια τάξη. Ελάχιστε αλλαγέ, ε, κάποιε προσαρμογέ. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε και θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι μπορούμε να θέλουμε να έχουμε μια οικονομική στρατηγική που θα βάλει την Ευρώπη προς τον δρόμο της ανταγωνιστικότητας να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί με ημίμετρα και με σταδιακές αλλαγές. Χρειάζεται να κινηθούμε γρήγορα. Πρέπει να δούμε ότι οι συνήθεις ρυθμοί δεν θα προστεύσουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, δεν θα προασπιστούν αυτές οι αλλαγές στα κοινωνικά μας μοντέλα, αντιθέτως μάλιστα Αυτά τα κοινωνικά μοντέλα θα κινδυνεύσουν εάν δεν προσαρμοστούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που δίνει περισσότερες προκλήσεις. Άρα χρειάζεται μια κοινή προσπάθεια. Πρέπει τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και η κοινωνία όλοι μαζί να κινηθούν. Και χρειάζεται και ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη του Κοινοβουλίου αυτού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να διαμορφωθεί η στρατηγική και για να προβάλλεται στον κόσμο αυτή η στρατηγική. Την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναφέρει ποια θα είναι τα βασικά στοιχεία στρατηγική που θα προταθεί επίσημα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα επικεντρώνεται επί τριών προτεραιοτήτων. Ευφυή ανάπτυξη, ενταξιακή ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη. Πρώτα απ' όλα, βασικό κινητή ανάπτυξη πρέπει να είναι η γνώση. Γνώση και καινοτομία που θα παράγει τι αυριανέ ιδέε, τι αυριανέ δεξιότητε, την αυριανή τεχνολογία. Δεύτερον, θα πρέπει να παραμείνει η ευρωπαϊκή, το κοινωνικό μοντέλο, να έχουμε περισσότερε απασχόλησει. Πρέπει να έχουμε υγιή, πλούσια, ασφαλή κοινωνία, όπου όλοι να αισθάνονται ότι μπορούν να παίξουν το ρόλο του. Αυτό σημαίνει ο κόσμο να έχει δουλειά και να αποκτά δεξιότητες και να εξαλειφθεί το στίγμα της φτώχειας. Το πρόβλημα της φτώχειας δεν είναι μόνο ένα εθνικό πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα για το οποίο απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τέλος, η οικονομία, η κοινωνική οικονομία τη αγορά θα πρέπει να μπορεί να εκμεταλλεύει τις ευκαιρίε τις μελλοντικέ. Μιλάω για βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να αναγνωριστεί η επιτακτική ανάγκη, η αλλαγή του κλίματο, να ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να αναγνωριστεί η πίεση που ασκείται στους πόρου. Και θέλουμε η ανταγωνιστική οικονομία να δημιουργεί νέε συνθήκε εργασία και για επενδύσει κυρίω για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, μια ευρωπαϊκή οικονομία που θα μπορεί να στέκεται σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Αυτές οι προτεραιότητες δεν είναι άγνωστες, αλλά το ότι δεν καταφέραμε ακόμα να ελοπίσουμε τους στόχους αυτούς ε, τους κάνει ακόμα πιο σημαντικούς και όχι λιγότερο. Εκεί που χρειάζονται ριζικές αλλαγές δεν είναι στο τι χρειάζεται να καθορίσουμε τι χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά το πώ υλοποιούνται οι στόχοι και τι χρειάζεται πραγματικά στην πράξη για να πετύχουμε. Πρώτα απ' όλα η στρατηγική θα πρέπει να είναι ολιστική. Δεν μπορούμε να διαλέγουμε διάφορα στοιχεία και ο καθένα να μπορεί να κάνει τα εύκολα, αυτά που τον κάνουν αισθάνονται καλά και να αφήνουμε τα πραγματικά προβλήματα και τι προκλήσει στου άλλου. Ε, και υπάρχουν πολλά στοιχεία. Η ενιαία αγορά, η ολοκλήρωση ενιαία αγορά, η ποιότητα των φορολογικών μας συστημάτων, πώς δαπανώνται τα χρήματα σε καιρό εντατικών πιέσεων επί των δημοσιονομικών, για να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία. Δεύτερον, η στατική μας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Δεν θα μπορεί η ευρωπαϊκή κοινωνία να μπει στο δρόμο για το μέλλον εάν αυτό γίνεται εις βάρος με το, με το κόστος της δημιουργίας κοινωνικών συγκρούσεων. Θέλουμε να, έχουμε, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, να καταπολεμήσουμε το στίγμα, την κατάρα της φτώχειας, βασική στόχη. Γι' αυτό θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε τις χρηματοδοτικές αγορές, θέλουμε ισχυρό οικονομικό τομέα που να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και την έρευνα. Θα πρέπει να, να αντιμετωπιστούν οι ευθύνε που φέρουν κάποιοι έναντι κυβερνήσεων και κοινωνιών θα πρέπει η στρατηγική να δέχεται ότι η σωστή εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι κάτι αναγκαίο σήμερα. Τρίτον, δεν θα πρέπει να συγχαίουμε ένα γενικό όραμα για την ευρωπαϊκή οικονομία με το θέμα ποιος αναλαμβάνει τι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφισβήτηση αρμοδιοτήτων. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία μια Ευρωπαϊκή προσέγγιση. Είναι προφανέ στην περίοδο τη παγκοσμιοποίηση όταν πρέπει να συζητούμε με του Αμερικανού, με του κινέζου, με του Ρώσους και με άλλου, ότι η προστιθέμενη αξία μια κοινή προσεγγίσεω, Παραδείγματο χάρη του G20, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια Γαλλική Προεδρία από τον πρόεδρο τη Γαλλία και από μένα, που προτείναμε στον Αμερικανό πρόεδρο να αποδεχτεί αυτέ τι συνόδου κορυφή. Αυτή Τέτοιου είδου σύνοδοι είναι απαραίτητε για να γνωριστεί ότι μπορούμε να βασιζόμαστε πολύ περισσότερο να, μετράμε περισσότερο να κινούμεθα μαζί. Δεν έχει νόημα να αναγνωρίζουμε την παγκόσμια αλληλεξάρτηση και να αρνηθούμε την ευρωπαϊκή αλληλεξάρτηση. Γι' αυτό πρέπει να κινούμαστε μαζί. Πολλά πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο ακόμα βέβαια. Υπάρχουν εθνικέ ευθύνε. Ε, και αυτό περιμένουμε να κάνουν οι κυβερνήσει. Αλλά περιμένουμε κυβερνήσει να προσπαθήσουν πραγματικά να ακολουθήσουν και ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι κάτι απαραίτητο. Όχι για δώσουμε να εκχωρηθούν εξουσίες στις Βρυξέλλες. Δεν είναι αυτός ο στόχος, αλλά να βοηθήσουμε να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στις κοινωνίες μας, ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ευμάρεια και μεγαλύτερο καλό και θετικά στοιχεία για τους πολίτες μας. Θα πετύχουμε μόνο αν είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε, όχι δίπλα ένα στον άλλον και ο ένα εναντίον του άλλου. Άρα χρειάζομαστε ε, σαφή επιμερισμό των εθνών σε όλα τα επίπεδα και χρειάζεται σωστό συντονισμό στο οικονομικό επίπεδο. Η συνδείξη τη Αβώνα μα δίνει τα αναγκαία μέσα. Θα τα χρησιμοποιήσω τα εργαλεία αυτά. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λοιπόν, τι είδα σε αυτό που έγινε. Είδα ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα προβλήματα. Μπορώ να συγκρίνω τι συζητήσει που έγιναν τώρα με τι συζητήσει που είχαν γίνει πριν από πέντε χρόνια, όταν συζητούσαμε τη στρατηγική τη Λισαβόνα. Και μπορώ να σα πω Επιτρέψτε να σας πω ειλικρινά και ανοιχτά ότι είδα μεταξύ των αρχηγών και κρατών και κυβερνήσεων μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, επίγνωση της ανάγκης συνεργασίας και επίσης ποιοι εξωτερικοί περιορισμοί υπάρχουν σε αυτή την ευρωπαϊκή οικονομία. Πραγματικά ειλικρινά πιστεύω ότι αυτή τη φορά εθνικά συμφέροντα δεν θα αντισταθούν εκ νέου στην ανάγκη για στενότερο συντονισμό και αποτελεσματικό σύστημα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Επίσης, χρειάζονται σημαντικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμβολα, για να δείξουν πού πάμε, τι θα κάνουμε. Κάποια συγκεκριμένα σχέδια που θα προτείνουμε, προγράμματα, όπως σχέδιο για καινοτομία, για ένα νέο πρόγραμμα για τα σχολεία, σωστή βιομηχανική πολιτική, ψηφιακό πρόγραμμα, ψηφιακή ατζέντα, πράσινες τεχνολογίες και συγκεκριμένο σχέδιο ή δράση κατά της ένδυας. Προγράμματα που έχουν αξία και θα έχουν αντίκτυπο προγράμματα που δείχνουν γιατί η Ευρώπη δίνει κάποια κομμάτια της λύσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μιλά απλώς, δεν μένει στα λόγια, αλλά και δρά. Θα κλείσω καλώντας εσά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δείξετε ισχυρή υποστήριξη προς αυτά τα προγράμματα, σαν νομοθέτε, σαν δημοσιονομική αρχή, αρχή του προπολογισμού και σαν υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής δράσης σε κάθε γωνιά τη Ευρωπαϊκή Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα θα ακούσουμε εκ μέρους των πολιτικών ομάδων και πρώτα εκ μέρους του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Χριστιανών Δημοκρατών, ο κύριος Ζωζεύ Ντόλ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11 η Φεβρουαρίου ήταν το πρώτο που συγκροτήθηκε και στο οποίο προείδρευσε ο πρόεδρος Χέρμαν Βαν Ρομπόη, τον οποίο και καλωσορίζω και χαιρετίζω την πρώτη του παρουσία εδώ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Βαν η ομάδα του ΕΛΚΑ έχει υψηλέ προσδοκίες από εσά. Χαίρομαι για το ρεαλιστικό και θετικό πνεύμα που δείξατε από την ανάληψη των υποχρεώσεών σας. Αλλά περιμένω από εσά, αλλά και από το Συμβούλιο των Υπουργών, να αντιληφθείτε και να συνειδητοποιήσετε ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας οι σχέσεις σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αλλάξει χαρακτήρα και φύση. Είμαστε και εμείς πλέον αρμόδιοι για τις πολιτικές αποφάσεις, επίσης όρες με το Συμβούλιο. Και αυτό έχει όχι μόνο νομικές συνέπειες, αλλά και πολιτικές επιπτώσεις. Ας έρθουμε τώρα στην ουσία της συζήτησης 11 Φεβρουαρίου, που είναι κυρίως η στρατηγική του 2020, αλλά και το ευρώ και η οικονομική και η δημοσιονομική στρατηγική. Γιατί η κερδοσκοπία κατά του ελληνικού χρέους και του ευρώ ήταν καλά όλα αυτά και η αναπάντηχη καλεσμένη της βιβλιοθήκης του Σολβέ. Αλλά η αποδυνάμωση του κοινού νομίσματός μας οφείλεται μόνο στην ελληνική κρίση ή μήπως το ευρώ ε, υφίσταται τις άμεσες επιθέσεις εκείνων που δεν βλέπουν με καλό μάτι την ισχύ του και την ισχύ των ε, κρατών που το εφαρμόζουν. Δεύτερη ερώτηση. Θα πρέπει να περιμένουμε να επιδεινωθεί η κατάσταση σε ορισμένες χώρες της ζώνης ευρώ για να επέμβουμε, όπως συνέβη στην Ελλάδα. Η ΔΕΜΗ τι προβλέπετε για να διορθωθεί η αστοχή αβολή στις, πιο, στις χώρες που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Και αυτό σας ερωτώ, Πρόεδρε Βαν Ρομπόη. Και θέτω όλες αυτές τις ερωτήσεις, γιατί χαίρομαι μεν για τα μέτρα αλληλεγγύης που θεσπίστηκαν την 11η Φεβρουαρίου, αλλά έχω σοβαρότατες επιφυλάξεις για το γεγονός ότι εμείς οι Ευρωπαίοι βρισκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Και ποια είναι η περίσταση αυτή ε, ο ελληνικός συναγερμός μας έδειξε ότι θα πρέπει να λάβουμε τολμηρές αποφάσεις για να δώσουμε επιτέλους στο ευρώ την αξία του και, την, και να γίνει πολιτική έκφραση το κοινό μας νόμισμα. Γιατί μιλάμε για, για οικονομική διακυβέρνηση, για νομισματική διακυβέρνηση, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη πιο απλοί και να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί προγραμματίζοντας και θεσπίζοντας έναν γνήσιο δημοσιονομικό συντονισμό των χωρών μελών της Ζώνης Ευρώ. Ο Εντουάρ Μπαλαντούρ, ο πρώην Γάλλος Πρωθυπουργός, αναγνώρισε την ανάγκη ε, νέας εκχώρησης ε, τμήματων κυριαρχίας και δεν είναι εύκολο να το παραδεχτεί κάτι τέτοιο ένας Γάλλος. Δεν λέω ότι η εθνική ε, προπολογισμοί θα πρέπει να υποβάλλονται από το Ευρωγκρουπ πριν υποβληθούν στις, ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτή την τολμηρή ιδέα και θα ήθελα να την εξετάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να την αναλύσει πολύ σοβαρά. Με σωστό συντονισμό των προπολογισμών, οι χώρε ευρώ θα έχουν πολύ μεγαλύτερο βάρο και περιθώριο λιγμών και μάλιστα περιθώριο λιγμών άνευ προηγουμένου. Και αυτή η ισχύ θα του δώσει ακόμη μεγαλύτερο βάρο και αποφασιστική σημασία στο παγκόσμιο προσκήνιο. Βέβαια, κάτι τέτοιο προαπαιτεί συσπήρωση των ευρωπαϊκών δυνάμεων και στις διεθνείς ε, οικονομικές ε, οργανώσεις, όπου η Ευρώπη θα πρέπει να ε, εκφράζει ενιαία φωνή. Η περίπτωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκεί τα δικαιώματα ψήφου καθορίζονται ανάλογα με το οικονομικό βάρος των χωρών. Με τέτοια κριτήρια οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν 16,7%. 6% η Ιαπωνία, 3,6% η Κίνα και οι έξι ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18,49%. Αν όμως είχαμε ενιαίο μέτωπο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν 23% των ψήφων και όλες ε, οι ευρωπαϊκές χώρες 32% αν ήταν ενωμένε. 32% των ψήφων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που είναι σχεδόν το διπλάσιο της ισχύω των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η αλήθεια του συσχετισμού δυνάμεων στον κόσμο. Και ακριβώς επειδή υπάρχει διχασμός και διχόνοια, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει όλο, όλο το βάρο. Είναι παραδεκτό κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι είναι πια απαράδεκτο. Θα πρέπει οι χώρες του ευρώ να ανοίξουν τα μάτια τους μπροστά σε αυτές τις περιστάσεις και να δουν τι συμπεράσματα θα αντλήσουν. Γιατί πολύ συχνά, πολύ γρήγορα η ανάγκη θα τους υποχρεώσει να συσπηρωθούν και όχι να αγκιστρώνονται σε κάποιες επιφάσεις οικονομικής κυριαρχίας που είναι κάποια επικίνδυνα προσχήματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε του ΕΛΚ. Εκ μέρου ε, τη Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το λόγο έχει ο κύριο Στίβεν Χιούζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Πρόεδροι. Από την αρχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης έχουν προσταθεί πολλά εκατομμύρια στους ανέργους της Ευρώπης και μέχρι τα τέλη του χρόνου πάνω από 25 εκατομμύρια άτομα θα είναι χωρίς ε, δουλειά. Αυτά που προσπαθήσαμε να πετύχουμε το δεκαετία του 90 έχουν καταστραφεί τα τελευταία δύο χρόνια και παρά τις προσπάθειές μας ε, το σύστημα απαιτείται με κατάρρευση. Η οικονομική ανάπτυξη είναι εξαιρετικά ασθενής και πολλοί ε, έχουν εκφράσει φόβους για το μέλλον των κοινωνιών μας. Και κάποια από τα κράτη-μέλη μας χρειάζονται πραγματικά απελπισμένα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη υπό τους όρους της ε, ε, τεράστιας κερδοσκοπίας. Αυτό είναι το ζωφερό οποίο στο οποίο η Ευρώπη πρέπει να επαναεφεύρει το μέλλον της με την κοινωνική και περαιτέρω ανάπτυξη. Κύριε Μπαρόσο, Πού θέλουμε να οδεύσει η Ευρώπη μέχρι το 2020. Πολύ σημαντικό ερώτημα, αλλά μπορούμε πραγματικά να ασχοληθούμε με τόσο μακρινό μέλλον χωρίς να κοιτάξουμε τι γίνεται τώρα με τους πολίτες μας που πλήττονται από την κρίση, που αναρωτιούνται τι θα κάνω αύριο, θα έχω δουλειά, θα έχω δυνατότητα να βρω μια καινούργια δουλειά. Τι απάντηση θα τους δώσουμε. Δεν μπορώ να γυρίσω αύριο και να πω στην περιφέρειά μου και να πω στον κόσμο ότι ε, κοιτάξτε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, έχουμε ένα σχέδιο για το 2020 τη στιγμή που δεν έχω απάντηση να δώσω για το τι θα κάνουν αύριο, αν θα έχουν μια εξαπρεπή δουλειά, με εξαπρεπή μισθό. Το Δεκέμβριο τέθηκε ένα τέτοιο θέμα από το Συμβούλιο. Μέχρι το 2011 τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, ενισχύσουν, να ενοποιήσουν ε, τις ε, δημόσιες δαπάνες τους. Αλλά παράλληλα θα υπάρχει πολύ μικρή ανάπτυξη και έτσι δεν θα μειωθεί η ανεργία. Και αυτό θα πλήξει ιδιαίτερα τους πιο ασθενείς ομάδες. Πρόεδρε Φαρόμπα και Πρόεδρε ε, Μπαρόσο να σκεφτείτε την ε, επωνομαζόμενη στρατηγική εξόδου. Θα πρέπει να βρούμε έναν ανθρώπινο τρόπο, έναν ηθικά υπεύθυνο τρόπο να εξέλθουμε από την κρίση και σε οικονομικούς όρους. Και αυτό δεν θα το πετύχουμε αν επικεντρωθούμε μόνο σε μακροοικονομικούς όρους σε ό,τι αφορά την γρήγορη ενοποίηση. Θα πρέπει να γίνει πραγματικά κοινωνική ε, ενίσχυση και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν μόνο μέσω των, με οικονομικούς όρους. Για να μην καταστούν και οι, μακροπρόθεσμα, οι προσωρινά άνεργοι μακροπρόθεσμα άνεργοι. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταστρώσουμε μια στρατηγική εισόδου στην σύγχρονη αγορά και θα πρέπει να καθορίσουμε έτσι τον χάρτη του πορείας μας μέχρι το 2020 σε ό,τι αφορά τις διατρατικές πολιτικές, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό τομέα για να δημιουργηθούν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια καινούργιε θέσει εργασία μέχρι το 2015. Θα πρέπει σαφέστατα να δηλώσει στο Ερνό Συμβούλιο το Συμβούλιο α, τις θέσεις τους και πέρα από τις αστυνομικές ε, ιδιότητες του Συμφώνου Σταθερότητας χρειάζονται πολλά παραπάνω. Θα πρέπει φυσικά οι δημόσιες δαπάνες να παραμείνουν σε τομείς ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Αυτό θα απαιτήσει και ε, ένα άλμα στην σε ό,τι αφορά την οικονομία και θα πρέπει να δοθεί εντολή στον Πρόεδρο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταρτιστεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το Δεκέμβριο του 2010. Κύριε Φανρόμπα και κύριε Μπαρόσο, ε, θα πρέπει να αμφισβητήσουμε κάποια από τα δεδομένα τα οποία είχαμε ως τώρα, αν θέλουμε να αλλάξουμε την ιστορία αυτή και αν θέλουμε να διδαχτούμε από την κρίση. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν η στρατηγική του 2020 αφορά τον άνθρωπο, τις θέσεις εργασίας, αν ενσωματέσει μια φιλόδοξη ατζέντα για τις ε, θέσεις εργασίας σας. Καλό να κάνετε ό,τι μπορείτε για να βάλετε τον άνθρωπο, τον πιο ευάλωτο άνθρωπο στον πυρήνα του Ευρωπαϊκού Project. Σας ευχαριστούμε κύριε Χιούς. Από την ομάδα των φιλελευθέρων τώρα θα εκφωνήσει ομιλία ο πρόεδρος της, ο κύριος Γκίβερ Χόφστατ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να περάσουμε στο πιο α, κατεπήγον πρόβλημα, γιατί μπορούμε να μιλάμε για το 2020, αλλά έχουμε ένα κατεπήγον πρόβλημα σήμερα, την Ευρωζώνη, την Ελλάδα, και θα πρέπει να εξεύρουμε λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Νομίζω ότι καταρχάς κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να αναλάβει το Κοινοβούλιο πρωτοβουλία στον τομέα αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε τι έγινε ακριβώς στην Ελλάδα. Γιατί σήμερα λάβαμε αντιφατικές πληροφορίες. Η Ελλάδα δηλώνει ότι έδωσε και διαβίβασε όλες τις πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκ παραλλήλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Eurostat δηλώνει ότι όχι, δεν λάβαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Εκ παραλλήλου, οι τράπεζε επενδύσεων, Goldman Sachs, ε, Stanley, Deutsche Bank, ε, ελαχιστοποιούν το δικό τους ρόλο στην ε, υπόθεση της Ελλάδας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καθήκον του Κοινοβουλίου μας, Πρόεδρε, να διοργανώσουμε το συντομότερο δυνατόν με τις αρμόδιες επιτροπές ακροάσεις για τα θέματα αυτά, ακροάσεις των αρμόδιων φορέων, να μάθουμε τι ακριβώς έγινε στην περίπτωση της Ελλάδας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για διευθυντικά μέτρα, για λύσεις, για μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν καταρχάς δεν έχουμε καθορίσει τι έγινε όντως το 2008, το 2009 και πιο πριν στην υπόθεση της Ελλάδας και νομίζω ότι είναι απόλυτα απαραίτητα, απαραίτητο να ακούσουμε όλες τις πλευρές. Κατά δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ελληνικού χρέους. Μία λύση υπάρχει νομίζω η οποία είναι δέουσα. Διάβασα χτες ε, το άρθρο του κ. Σόρος στους Financial Times σχετικά με το θέμα αυτό και του Γιώσκα Φίσερ πριν από κάποιες ημέρες ε, στο γερμανικό τύπο, ο οποίος ε, αναφέρει αυτό που πολλοί αναφέρουν, ότι η καλύτερη λύση για την το ευρωπαϊκό χρέος είναι μια ευρωπαϊκή λύση. Ευρωπαϊκά ομόλογα του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου χωρίς κόστος για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, αλλά με μια λύση για το μέλλον. Και νομίζω ότι είναι και καθήκον του Κοινοβουλίου μας να ζητήσει από το Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο, να σκεφτούν να αναλογιστούν αυτή τη λύση. Να περάσουν και να υπερβούν τα εθνικά συμφέροντα των ε, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλογιστούν αυτή τη δυνατότητα. Και κατά τρίτον πρόεδρε, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό τμήμα της συζήτησης αυτής είναι το τι θα κάνουμε για το 2020. Η Ελλάδα είναι εξαιρετικό παράδειγμα για το τι πήγε στραβά σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ήταν υπερβολικά αδύναμη και το κενό, το χάσμα μεταξύ ε, γερμανικής και ελληνικής ε, οικονομίας ε, οξύνθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια, δεν μειώθηκε. Γιατί θα πρέπει λοιπόν η, το Συμβούλιο και η Επιτροπή να αναγνωρίσουν ότι ο ανοιχτός τρόπος συντονισμού δεν ήταν καλή λύση. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο εργαλείο στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πιο τολμηρό εργαλείο είναι η οικονομική διακυβέρνηση στο ιστορικό της Ένωσης. Ελπίζω, κύριε Μπαρόσο, σε λίγες ημέρες, στις αρχές Μαρτίου, στο τέλη Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, να α, μας παρουσιάσετε σχετικό έγγραφο. Και ελπίζω τα συμπεράσματα να συμπεριληφθούν τα συμπεράσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι είναι το αποτέλεσμα, διακυβερνητική ανεκτή μέθοδο συντονισμού, λίγο πιο γρήγορη, λίγο βελτιωμένη, λίγο πιο γρήγορη, αλλά παραμένει διακυβερνητική αυτό που σας δούμε είναι να ηγηθείτε, να ηγηθείτε σε αυτή την οικονομική πολιτική, σε αυτή την οικονομική διαβίρυνση μαζί με τον Όλη Ρεν, να μας υποβάλλετε μια τολμηρή πρόταση για οικονομική διακυβέρνηση στο ιστορικό της Ένωσης, γιατί είναι ανοησία, ανοησία να υπάρχει νομισματική ένωση αφενός και να μην υπάρχει αφετέρου ε, οικονομική πολιτική και οικονομική ένωση και αυτό το καταδεικνύει το παράδειγμα της Ελλάδας. Έχει έρθει λοιπόν ο καιρός, ε, συνάδελφοι, να λάβουμε κάτι πιο τολμηρό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω στις 3 Μαρτίου να είναι πολύ πιο φιλόδοξες οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Θα, θα θέλετε να απαντήσετε τώρα στις ε, ερωτήσεις από τις μπλε κάρτες. Μία γαλάζια κάρτα βλέπω εδώ. Κύριε Βαρχόστατ, τι λέτε ότι οι χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη θα πρέπει να γλιτώσουν χώρες που είναι στην Ευρωζώνη, να τις βοηθήσουν. Αυτό προτείνεται. Απάντηση του κυρίου Βερχόφστατ εκτός μικροφώνου. Ίσως το εγγύς μέλλον θα πρέπει να βοηθήσουμε τη Βρετανία, διότι βλέπω και το φορολογικό έλλειμμα, το οικονομικό έλλειμμα της Βρετανίας που είναι μεγαλύτερο από το οικονομικό έλλειμμα της Ελλάδας. Οπότε ίσως χρειαστεί να βοηθήσουμε τη Βρετανία. 12,9% του ΑΕΠ περίπου είναι το οικονομικό έλλειμμα αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε αξιόπιστη, αξιόπιστη στρατηγική προς την Ευρωζώνη. Και είμαι βέβαιος, ίσως όχι αύριο αλλά μεθαύριο, θα έρθει η στιγμή όπου και η Βρετανία θα γίνει μέλος της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ η πρόεδρος Ρεμπέκα Χάρμς από τους Πράσινους και την Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Η πρόεδρος των Πρασίνων, η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ αξιότιμοι πρόεδροι, ελπίζω το Βρετανικό νηπιαγωγείο να ειδέμισε για να μπορέσουμε να συντηρηθούμε και πάλι. Θα ήθελα να ξεκινήσω να μιλάω για την Ευρώπη του 2020 και μετά να συνεχίσω ε, με το θέμα της Ελλάδας. Αλλά επειδή παρενέβη και η δεξιά πλευρά του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να πω ότι αυτό που θεωρώ ότι βοηθάει το λιγότερο στην όλη ε, κατάσταση με την Ελλάδα είναι η μια στάση κατά της Ελλάδας, μια εθνικιστική στάση, μια αντιευρωπαϊκή στάση. Αυτό βοηθάει το λιγότερο από όλα. Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό που κατέστησε σαφές στην κρίση, τονίζεται ιδιαίτερα σήμερα, είναι σφάλματα τα οποία γίνονται εδώ και καιρό και θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Φερχόφστατ. Αν δεν θέλουμε να διαδραματιστούν, να εξελιχθούν αντιευρωπαϊκές τάσεις, θα πρέπει να συζητήσουμε ποιος στις Βρυξέλλες έχει ευθύνη για το γεγονός ότι επί σειρά ετών, κατά πάσα πιθανότητα σε όλη την προετοιμασία της Ευρωζώνης, μπόρεσαν να κρυφτούν τόσα πολλά πράγματα στην Ελλάδα και νομίζω ότι κύριε Μπαρόσο έχετε σημαντική ευθύνη. Αυτό θα πρέπει να αποκαλύψετε γιατί όσο του το αποκαλύψουμε αυτό θα βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου σε ό,τι αφορά τις ευθύνε. Και κατά δεύτερον και στην Ελλάδα φυσικά θα πρέπει να αλλάξουν πολλά. Αυτό είναι μια φιλική, αν θέλετε, αντιμετώπιση της Ελλάδας στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Αν η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κληθεί να συνδράμει, το οποίο δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να αποκλείσω, θα πρέπει πραγματικά οι Έλληνες κάτι να αλλάξουν σε ό,τι αφορά τον τεράστιο αυτό δημόσιο κλάδο. Νομίζω ότι από ό,τι μου έχουν πει οι Έλληνε με του οποίου έχω μιλήσει, 25% απασχολείται στο δημόσιο τομέα. Και αυτό είναι καλό γιατί έχουν ήδη προετοιμαστεί ε, αλλαγέ. Αλλά θα πρέπει να αλλάξει κάτι και στι δαπάνε αλλά και στα εισοδήματα. Και θεωρώ ότι ο κύριος Πανδρέου με την ιδέα του σε ό,τι αφορά την φορολογική δήλωση των υψηλών μισθολογικών ε, κλιμακίων ε, έχει καλές ιδέες. Δεν νομίζω. Αυτό μάλλον θα φωτίσει καλύτερα το πόσο μπορεί να βελτιωθεί η πλευρά των προσόδων στην Ελλάδα με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Για να πληρώνουν φόρους και αυτοί που ζουν πλούσια στην Ελλάδα. Θα μιλήσετε αργότερα, φαντάζομαι, για τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Αλλά θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη στρατηγική για το 2020. Κύριε Μπαρόσο, δεν μιλήσατε καθόλου για τις αποτυχίες της στρατηγικής τη Λισαβόνας και νομίζω ότι η έλλειψη, αν θέλετε, η απουσία αξιολόγησης της συνθήκης της Λισαβόνας αποτελεί κακό ιονό για την ε, επιτυχία της νέας στρατηγικής, η οποία δεν είναι κατ' ουσία αρνητική. Κλείνει το μικρόφωνο της ομιλητριάς. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο σας γιατί είναι αδύνατο να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας αν ο καθένας συστηματικά υπερβαίνει το χρόνο. Το κύριο Σκύρκοπ. Πρόεδρε, καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Βερχοφστάτ που μας υπενθύμησε το πώς απέτυχε η οικονομική πολιτική της αριστερά στην, στον Αμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή κύριε Βερχοφστάτ και ελπίζω συναδελφοί μου και εγώ να μπορέσουμε να το διορθώσουμε αυτό στις επικείμενες γενικές εκλογές. Πρόεδροι, πριν ακόμα την πρόσφατη κρίση, οι οικονομίε τη Ευρώπη ε, έχαναν έδαφο έναν των μεγάλων αντιπάλων μα και ανταγωνιστών μα. Το επίπεδο ανάπτυξη ήταν λιγότερο και υψηλότερη ανεργία και η θέση μα όσον αφορά το εμπόριο επιδεινωνόταν και το μερίδιο όμω όσον αφορά την παραγωγή, την παγκόσμια μειωνόταν. Ξεκινήσαμε τη στρατηγική τη χωρί να έχουμε αρκετέ δεσμεύσει και πειθό και δεν πέτυχε και αυτό δεν μας εκπλήσει. Η Ευρώπη του 2020 δεν πρέπει να ακολουθεί στον ίδιο δρόμο και χαίρομαι που η ομάδα μου ήταν μεταξύ των πρώτων που υπέβαλαν προτάσεις για να επιτευχθεί πρόοδος σε αυτή την πορεία. Χρειάζεται νέα πορεία τη οικονομία μας. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι κυβερνήσεις δεν δημιουργούν παραγωγικές θέσεις απασχόλησης, ούτε αυξάνουν το επίπεδο διαβίωση, Μόνο οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και επιτυχείς επιχειρηματίες μπορούν να το κάνουν αυτό. Τα κράτη-μέλη μας και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να τους υποστηρίξουν αυτούς μειώνοντας το άχθος που αντιμετωπίζουν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να έχουμε μια δυναμική οικονομία αν κάνουμε, έχουμε μεγαλύτερε απαιτήσει από εκείνου που δημιουργούν ανάπτυξη και θέσει απασχόληση με επιβάρυνση φορολογική και γραφειοκρατικού κανόνε. Θα πρέπει να θαρρύνουμε περισσότερη ανάπτυξη και έρευνα, να βελτιώσουμε την ανώτατη εκπαίδευση και καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση, όπω είπε μόλι τώρα ο κύριο Μπαρόζο, ο πρόεδρο Μπαρόζο. Η εσωτερική αγορά θα πρέπει να ζωγονηθεί και να επεκταθεί σε νέου τομεί. Πρόεδροι, τα, οι προκλήσει είναι πάρα πολύ μεγάλε. Επί τρει αιώνε, οι πιο ισχυρέ οικονομικέ δυνάμει στον κόσμο ήταν εκείνε που ήταν οι πιο φιλελεύθερε και πιο δημοκρατικέ, που είχαν το δημοκρατικότερο σύνταγμα. Η ελευθερία και η οικονομική ευμάρεια προχωρούσαν χέρι με χέρι. Μπαίνουμε σε νέα εποχή, αλλά το τέλο, αυτού του αιώνα Μεγάλε η οικονομική ισχύ μπορεί να πήγε σε χώρε που είχαν μη δημοκρατικέ ε, κυβερνήσει. Αυτό ο αυταρχικός καπιταλισμό δεν μπορεί να συγκριθεί, να ανταγωνιστεί κανονικά με το δημοκρατικό καπιταλισμό που έχουμε. Ελπίζουμε τα κάτι αυτά να απελευθερωθούν, να μπορούμε να του δώσουμε ενθαρρύνσει, αλλά ξέρουμε του κινδύνου. Είναι λοιπόν προ όφελο των πολιτών να δημιουργήσει το πρόγραμμα το 2020 ε, καλέ θέσει απασχόληση και βελτίωση του επίπεδου διαβίωση. Και προ όφελο του ελεύθερου κόσμου το πρόγραμμα για το 2020 να οδηγήσει σε ένα ισχυρότερο οικονομικό μέλλον για του πολίτε μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λόταρ Μπίσκι από την ΚΟΕ και τη Σκανδιναβική Αριστερά. Κύριε Πρόεδρε, μια παροιμία λέει ότι στην ανάγκη φαίνεται ο φίλος. 27 κυβερνήσεις υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε μία προσπαθεί με τον τρόπο της να σώσει τις μεγάλες βιομηχανίες και τις τράπεζές της. Αυτό τι σημαίνει. Ως τώρα αυτό σήμαινε πιο πολλά χρέη από αυτά που αναλογούσαν σε κάθε κράτος και λιτότητα, μεγάλη λιτότητα. Εφημιστικά το αναφέραμε αυτό ως ε, ιδιωτικοποίηση του κινδύνου ζωής, ε, μείωση της, ε, των μισθών και το καθεξής. Με τα πακέτα αυτά για τις τράπεζες κερδοσκοπούν τώρα αυτές ακριβώς κατά των κρατικών προϋπολογισμών γιατί οι τράπεζες έχουν περάσει παραπέρα από τα κράτη. Έχουν σωθεί με δισεκατομμύρια η Hypo Bank για παράδειγμα στην ε, Γερμανία και τώρα παίζουν με την Ελλάδα. Κερδοσκοπούν με τα χρήματα του έντιμου φορολογούμενου που δεν έχει ε, λογαριασμό στην Ελβετία. Και δεν χαίρομαι καθόλου να χρησιμοποιώ, συνάδελφε, αρνητικά γερμανικά παραδείγματα, αλλά στη Γερμανία ένα κόμμα ζητάει φορολογική ελάφρυνση και εκ παραλίλου καλούμε στην ελληνική κυβέρνηση να επιβάλλει επιπλέον φόρους. Αλλά εγώ πολύ φοβάμαι ότι τελικά αυτοί που θα πληρώσουν είναι εκείνοι που θα τα βγάζουν πέρα με το μισθό τους ήδη σήμερα. Και είναι παγκόσμιο εξαγωγέας ε, η Γερμανία, η Γερμανία που αποσύνδεσε εδώ και χρόνια το ύψος του μισθού από την παραγωγή, με κοινωνικό dumping. Η κρίση σημαίνει ότι έχουμε και την ευκαιρία, τη δυνατότητα να αλλάξουμε, να σημειώσουμε ένα σημείο καμπής, ε, να δημιουργηθούν ε, ελάχιστοι μισθοί για κάθε χώρο εργασίας. Θέλουμε κοινοτική εναρμόνιση των φόρων, αλλά κυρίως θέλουμε μια κοινή ρύθμιση και έλεγχο των χρηματοοικονομικών αγορών και πραγματικά κοινή αλληλέγγυα πολιτική, οικονομική και χρηματοοικονομική, δημοσιονομική. Και αυτή θα πρέπει να έχει δεσμευτικούς στόχους σε ό,τι αφορά και το περιβάλλον αλλά και την κοινωνική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Νάιτζελ Φαράζ, ο πρόεδρος ε, της Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Πρόεδρε τη Ευρώπη, περιμέναμε επί πολύ αυτή την ημέρα. Μα λέγανε ότι θα έχουμε πρόεδρο, θα έχουμε μια γενία, μια γενναία τεράστια, ένα γίγαντα πολιτικό. Τον άντρα που θα, πολιτι... θα ηγηθεί 500 εκατομμυρίων πολιτών, που θα εκπροσωπεί όλου μα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Τον άντρα που η δουλειά του τόσο σημαντική που βεβαίω θα πληρωνόταν περισσότερο από τον πρόεδρο Ομπάμα. Αλλά φοβούμαι ότι αυτό που πήραμε, εσά πήραμε. Και λυπούμε. Αλλά μετά από αυτή την επίδοση που μας, του λόγου σας, τι να πω, δεν θέλω να είμαι αλλά πώς να το πω, ε, έχετε το, το χάρισμα σαν να είσαστε πατσαβούρα και φαινόσαστε σαν υπαλληλίσκος τράπεζας εμφάνιση. Και το ερώτημα που έχω να θέσω, και όλοι μας διερωτώμεθα, ποιος είσαστε εσείς, δεν σας έχω ξανακούσει ποτέ, κανείς στην Ευρώπη δεν σας άκουσε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Πρόεδρε, Ποιος σας ψήφισε και τι μηχανισμό Ξέρω, δημοκρατία δεν είναι δημοφιλής για σας, όλους σας. Τι μηχανισμό χρησιμοποίησαν οι λαοί της Ευρώπης για να σας βγάλουν από τη θέση σας. Αυτό είναι ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αισθάνομαι, αισθάνομαι όμως ότι είστε ικανός και επικίνδυνος και δεν έχω αμφιβολία ότι έχετε πρόθεση να είστε ήσυχο δολοφόνος της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών κρατών εθνών. Φαίνεται να μισείτε την έννοια της ύπαρξης των εθνών κρατών, των εθνικών κρατών. Ίσως γιατί κατάγεστα το Βέλγιο, που το Βέλγιο είναι μη χώρα, λίγο πολύ. Αλλά εφόσον πήρατε αυτή τη θέση και αναλάβατε, τι είδαμε. Η Ελλάδα να γίνει προτεκτοράτο και τίποτα παραπάνω. Κύριε, δεν έχετε καμία νομιμότητα σε αυτή τη θέση, σε αυτή τη δουλειά. Και λέω με κάθε πεποίθηση, μιλώντα εκ μέρου τη πλειοψηφία των Βρετανών, όταν λέω ότι δεν σα γνωρίζουμε, δεν σα θέλουμε και όσο πιο γρήγορα σα διώξουν, τόσο το καλύτερο. Well, as you said, Mr. President... Όπως είπατε, δεν θέλετε καθόλου να είστε αγενείς. Ευτυχώς που το είπατε. Προτιμώ αυτή σας μόνο τη δήλωση να κρατήσω, ότι δεν θέλατε να είστε αναγενείς. Μπελέ κάρτα από τον κύριο Ντόλ. Κύριε Φαράζ, συμφωνείτε να εφαρμόσουμε το άρθρο 9 της συνθήκης. Να ζητήσουμε έξοδο από την Ευρώπη, να φύγετε από την Ευρώπη και να ησυχάσουμε όλοι. Yeah. Okay, thank you. Ωραία, σας ευχαριστώ. Τι θέλετε. Διαδικαστικό. Διαδικαστικό ο κύριος Σούλτς. Εκτός μικροφώνου. Πολύ με παγωτεύετε, κύριε Πρόεδρε Μπούζεκ. Δεν είναι αποδεκτό, είναι παράδεκτο εδώ στο Κοινοβούλιο αυτό ένας πρόεδρος ομάδας να μιλάει έτσι ε, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να τον ε, από το καλή πατσαβούρα, όχι να του κάνει πολιτική κριτική δηλαδή. Και κύριε Πρόεδρε, αναμένω από εσά να κάνετε, να θίξετε θέμα διαδικαστικό. Δεν είναι τον αυτός ο άνδρας να καταπατάει την αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου και να πω στον πρόεδρο ε, Ντόιλ το θέμα δεν είναι να βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως καλύτερα θα ήταν ο κύριος Φαράζ να δώσει την έντρα του άμα τόσο πια τον δυσαρεστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Όπως είπα και πριν στον κύριο πρόεδρο Φαράζ πριν από δύο μήνες, σαν σήμερα καλή ώρα, τέτοιου είδους ομιλίες που ασκούν προσωπική επίθεση κατά συγκεκριμένο προσώπου είναι απαράδεκτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είχα σχετική συζήτηση με το θέμα αυτό, για το θέμα αυτό με τον κύριο Φαράς και του είχα επιστήσει την προσοχή στο θέμα αυτό. Δεν απαγορεύονται οι, εθνικές, οι προσωπικές επιθέσεις. Αυτή είναι η δική μου θέση. Είναι εκτός μικροφώνου ο κύριος Φάρατζ. Τι είναι προσωπική δήλωση, κύριε Φαράζ. Ξέρετε, ίσως να μην σας αρέσουν αυτά που είπα. Αλλά σκεφτείτε τη δική σας συμπεριφορά. Εσείς μετά το δημοψήφισμα της Ιρλανδίας που οι Ιρλανδοί είπαν όχι, είπατε ότι η ομάδα μας με την υποστηρίζοντας το όχι άνοιξε την πόρτα στο φασισμό Είπατε ότι είχαμε συμπεριφερθεί σαν ομάδα στο Κοινοβούλιο, σαν το Χίτλερ και τους Ναζί στο Reichstag. Μας απόκριψε ο Ντάνι Κομπέτ ε, πνευματικά δύναμη, καθυστερημένη. Δεν μπορεί να τα έχετε όλα. Δεν ήταν προσωπική δήλωση αυτή κύριε Φαράς. Κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν προσωπική αυτή η δήλωση. Συγγνώμη, αλλά δεν ήταν προσωπική δήλωση. Θα πρέπει να τηρήσουμε τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την τάξη στη συζήτηση, παρακαλώ. Επόμενο Επόμενος ο είναι ο κύριος Φρανκ Βανέκε, από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να διαπιστώσω ότι η συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, γίνεται στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο σε μια χώρα την οποία μπορούμε να περιγράψουμε στο οικονομικό υπόβαθρο ως ε, την Ελλάδα της Βόρειας Θάλασσας. Γιατί όπως η Ελλάδα και το Βέλγιο μετά την Ιταλία και την Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος. Και αυτό το οφείλουμε σε έναν από τους προηγούμενους ομιλητές, τον πρώην Πρωθυπουργό Φερχόφστατ ο οποίος ε, με την τεχνητή παρουσίαση των προϋπολογισμών ε, μας έχει καταστρέψει. Ας μην ε, υποκρινόμαστε ότι μπορούμε να απαλύνουμε την κρίση με τη δημιουργία επιπλέον δημόσιου χρέους. Με ένα χρέος το οποίο κάποιος θα κληθεί να πληρώσει τελικά. Ήταν αυτές οι ευρωπαϊκές αποφάσεις οι οποίες μας οδήγησαν τελικά στην κρίση. Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις για τα κρατήρια του Μάστρετ, για το σύμφωνο σταθερότητας και η ίδια ευρωκρατική, αν θέλετε, στενομυαλά, στενομυαλιά, μας ε, χώνει στο σβέρκο την Τουρκία και μας κάνει να αγνοούμε τις γεωγραφικές πραγματικότητες και καλεί τον Ευρωπαίο, πολίτη να καταβάλει τεράστιο κόστος για μια χώρα που δεν είναι καν ευρωπαϊκή. Η λύση λοιπόν είναι η εθνική αρμοδιότητα, όχι η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Ευχαριστώ. Οι υπόλοιποι ομιλητέ. Η κυρία Κόριν Βόρτμαν Κόλ για δύο λεπτά. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε Μπούζεκ, Μπαρόσο και Πρόεδρε Φαρόμπαϊ. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαιρόμαστε όλοι που είσαστε εδώ σήμερα. Και δείχνετε με την έναρξή σας αυτή ότι θέλετε να δουλέψετε με φιλοδοξία, αλλά ακριβώς όπως προβλέπετε και ο ρόλος σας στη συνθήκη της Λισαβόνας και σας τιμάει αυτό. Είναι σημαντικό για το γεγονό ότι βρίσκεται εδώ πέρα για την ε, επερχόμενη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, που θα είναι σημαντική για το μέλλον τη Ένωση. Πρόεδρε και Πρόεδρε Μπαρόσο, ξέρετε ποιε είναι οι προτεραιότητε. Η πράσινη ε, οικονομία τη αγορά είναι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων και μιλάμε κυρίω για μικρομεσαίες επιχειρήσει που αποτελούν τον κινητήρα της απασχόλησης. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να λάβουν νέα όθηση και δεν μιλάμε μόνο για το εμπόριο και τις υπηρεσίες, μιλάμε και για την ευρωπαϊκή βιομηχανή μας. Θα πρέπει να καταστεί εκ νέου ανταγωνιστική. Και μιλάμε και για τον αγροτικό μας τομέα που θα πρέπει να είναι ποιοτικό σε ό,τι αφορά την παραγωγή των τροφίμων, που και αυτά θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και χρειαζόμαστε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να είναι πλούσιε σε γνώση, καινοτομία, βιώσιμη τεχνολογία. Αλλά η στρατηγική για το 2020 θα πρέπει να βασίζεται σε ένα γερό θεμέλιο. Και το γερό θεμέλιο τι σημαίνει, μια στρατηγική εξόδου η οποία θα συνδέεται με ένα ε, καλό πακέτο ανάπτυξης και σταθερότητες και ένα καλό πρόγραμμα ε, δαπανών στα κράτη-μέλη. Πρόεδρε, η παλιά συνθήκη της Λισαβόνας είχε πάρα πολλές ασαφείς ε, στοχοθετήσεις. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτώ, πώς θα ε, επιβάλλετε δεσμευτικές, δεσμευτικούς στόχους στα κράτη-μέλη εντός φυσικά των ορίων της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά τη διάσταση της επικουρικότητας. Σας ευχαριστούμε κυρία Βόρτμαν Κολ. Το λόγο έχει η κυρία Μαρίτα Σκοκ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με βάση τα στοιχεία που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 80, 80 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών διαβιούν ε, στο κατόφλι της φτώχειας. Αυτό είναι απαράδεκτο και μάλιστα εμποδίζει την απρόσκοπτη πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά έρχεται ο κύριος Φαρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας προσβάλλει κατάμουτρα ενώ η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια κρίση. Νομίζω ότι τέτοιου είδου άνθρωποι δεν έχουν θέση στην Ολομέλεια τη επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να επιβληθούν κυρώσει για τόσο ανάρμοστε συμπεριφορέ. Έχουμε τώρα την πρόταση για μια νέα στρατηγική της Λισαβόνας που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020. Η κοινωνική συνοχή και η φόρος ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και της οικονομικής ανάπτυξης. Και φυσικά θα πρέπει να εξέλθουμε από την κρίση αυτή γιατί μόνο αν ξεπεράσουμε την κρίση θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Και χρειαζόμαστε και περισσότερους πόρους πολύ περισσότερους από αυτούς που προβλέπονται σήμερα για την έξοδο από την κρίση. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε μια νέα ε, συμφωνία φιλόδοξη για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης, ένα νέο Dream Deal. Επίσης ε, θα πρέπει να επενδύσουμε στην ε, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να πατάξουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό που σοβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στις διαβουλεύσεις και τους κοινωνικούς εταίρους όλο, και περισσότερο διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις ε, θεωρούν την, την δραστηριότητα των ε, συνδικάτων ως απειλητική για τη λειτουργία τους. Λάθος, θα πρέπει να εμποδίσουμε την ε, θέσπιση και έγκριση οδηγιών που δημιουργούν μισθολογικό ντάμπινγκ. Ευχαριστώ. Κυρία Έκ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στόχος του στόχου για το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να απελευθερωθεί το δυναμικό των Ευρωπαίων πολιτών. Πολύ συχνά λησμονούμε ότι οι στρατηγικέ μα για την ανάπτυξη εφαρμόζονται προ όφελο των πολιτών μα και για το μέλλον των παιδιών μα. Αναμφισβήτητα, η στατική τη απέτυχε όταν προσπάθησε να συμπεριλάβει τα πάντα με τόσο ευρύ πρόγραμμα χάσαμε το στόχο, την, τον εστιασμό μας και τις δυνατότητες να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που είχαν τεθεί. Για τη στρατηγική για το 2020, για να είναι πιο αποτελεσματική, η μορφή θα πρέπει να αλλάξει και να έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα πρέπει να στεστούν οι προσπάθειες επί συγκεκριμένων λίγων τομέων όπου τα διάφορα θεμελιώδη στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Σαν το μόνο άμεσα εκλεγόμενο σώμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και με πλήρης εξουσίες για συναπόφαση το Κοινοβούλιο θα έχει λόγο στον αφατιστική για το 2020 ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα και ανοιχτή προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα ήταν καλό να συμπεριλάβουν το Κοινοβούλιο στις εργασίες που γίνονται για τη διαμόρφωση στρατηγικής του 2020. Ανοιχτή προσέγγιση και διαφάνεια είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μια Ευρώπη των πολιτών και είναι βασικά στοιχεία για να αποφευχθούν κρίσει όσον αφορά τα δημοσιονομικά, όπω η κρίση που πλήττει χώρε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι δακτυλοδεικτούν την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν επίση και άλλα κράτη-μέλη τα οποία έχουν αποφύγει την βαθμολόγηση και έχουν ξεγελάσει την Ευρώπη στον αφορά τα ελλείμματά του και το κατάφεραν με τα δικά του οικονομικά στατιστικά στοιχεία. Η μέθοδο του ανοιχτού συντονισμού τελικά τι έγινε. Κλειστή συνωμοσία και ανοιχτή ταπείνωση. Πρέπει να θυμηθείτε ότι αυτό που αληθεύει για τους πολίτες αληθεύει και για τις κυβερνήσεις. Η ελευθερία συνεπάγεται και ευθύνε. Δεν θα πρέπει τώρα οι, κυβερνή, οι κυβερνήσεις να υπομισθούν ε, τις ευθύνε τους, διότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι και αυτά σοβαρά. Χρειάζεται σοβαρότητα. Ο κύριος Φίλιπ Λάμπερτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνώ με την ιδέα να περιοριστεί ο αριθμό των στόχων τη στρατηγική του 2020. Αρκεί να είναι φιλόδοξη αυτή η στόχοι, λίγη και φιλόδοξοι, για το οικολογικό μα αποτύπωμα για παράδειγμα και δεν περιορίζομαι μόνο στο κλίμα. Θα πρέπει να ξαναβρούμε το στόχο του μείον 20% που ούτω ή άλλω υστερεί των αναγκών μα. Ούτε το 30% δεν είναι φιλόδοξο. Επίση, θέλουμε φιλόδοξου στόχου για τον περιορισμό των ανισοτήτων. Να μειώσουμε κατά 50% μέχρι το 2020 τη φτώχεια στην Ευρώπη. Δεν είναι και πάρα πολύ φιλόδοξο αυτό. Επίση, θέλουμε φιλόδοξου στόχου για την παιδεία, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη. Φιλόδοξου στόχου για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Όλοι αυτοί οι στόχοι όμω θα πρέπει να είναι καταμετρήσιμοι, ποσοτικοποιημένοι και δεσμευτικοί. Δεν ξέρω τι σύστημα θα βρείτε, μπόνους μάλους, ε, ε, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξουμε αποτελέσματα. Και αυτά τα αποτελέσματα δεν πρόκειται να ελοπίσουμε αν μας λείπουν δύο συγκεκριμένα συστατικά. Μία ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και μάλιστα αυστηρή ρύθμιση. Γιατί είναι πολύ ανησυχητική εδώ η θέση του Συμβουλίου και αυτά που μα είπε ο κύριος Βαν Ρόμποϊ. Και όπω είπε ο κύριος Ντόλ, όντω θα πρέπει να έχουμε νέε εκχωρίστημάτων τιμάτων κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στο φορολογικό και δημοσιονομικό τομέα. Χωρί φορολογικό, φορολογική και δημοσιονομική σύγκληση δεν πρόκειται να επανισορροπήσουν τα οικονομικά των κρατών μελών. Επίση, το θέμα τη φορολογία των ε, χρηματοπιστωτικών και οικονομικών συναλλαγών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, η κυρία Σουίμπερν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Να πω ότι υποστηρίζω την κατεύθυνση τη στρατηγική για το 2020 Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω τώρα την εποχή τη οικονομική κρίσεω. Και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιαστεί επί τη συγκρίσιμου ε, ανταγωνιστικού και οικονομικού ωφέλου. Ε, και να συγκεντρωθούμε κυρίω στην έρευνα και ανάπτυξη, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή σε αυτό τον τομέα. Θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητε όσον αφορά την ολοκλήρωση ευρωπαϊκή ενιαία αγορά για υπηρεσίε και αγαθά. Και χρειάζεται φιλόδοξη προσέγγιση για μια ενιαία αγορά για καινοτομία έρευνα. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την έρευνα και την ανάπτυξη και στα πανεπιστήμια και στις ιδιωτικέ επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τόσο ώστε να είμαστε στην πρώτη γραμμή μιας νέας βιώσιμης βιομηχανίας και νέων βιώσιμων τεχνολογιών. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε όμως όσον αφορά την νομοθεσία που εξυπηρετεί στο να παρεμποδίζει αυτές τις αναπτυξιακές διαδικασίες. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη σχέση μεταξύ ιδιωτικού τομέα και πανεπιστημιακή έρευνα, και θα πρέπει να διευκολύνουμε τη μεταφορά τεχνογνωσία, ώστε να, δημιουργήσουν, να δημιουργηθούν επιχειρήσεις που δημιουργούν και ευμάρεια. Χρειάζεται οικονομική ανανέωση, αλλά θα πρέπει να μειωθεί και το ε, διοικητικό άκτο κυρίως για τις μικροεπιχειρήσεις και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θα πρέπει οι οι δημόσιοι διαγωνισμοί να διευκολύνουν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να συμμετάσχουν και πρέπει να υπάρχει συνεργασία ε, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και πρέπει να ενθαρρύνουμε την καινοτομία σε όλου του τομεί. Ο κύριο Νικόλα Χουντή έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σήμερα στην Ελλάδα γίνονται μεγάλε απεργιακέ κινητοποίησει από του εργαζόμενου στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα έχει βγει στους δρόμους ο θυμός και η αγανάκτηση των εργαζόμενων απέναντι στα σκληρά μέτρα που παίρνει η ελληνική κυβέρνηση με την προτροπή της ευρωπαϊκής ένωσης ιδιαίτερα του τελευταίου πρόσφατου ευρωπαϊκού συμβουλίου όπου αντί σε αυτό το ευρωπαϊκό συμβούλιο να ληφθούν μέτρα υπέρ των αδύναμων οικονομιών να πάρθουν μέτρα για να τεθεί ένα τέρμα στους κερδοσκόπους αντί να δημιουργηθεί μια ομπρέλα οικονομική και κοινωνική αλληλεγγύη αντί να παραδεχτείτε ότι το σύμφωνο σταθερότητα δεν υφίσταται και η επαναφορά του θα φέρει μεγαλύτερη ύφεση αντί να παραδεχτείτε ότι η συνθήκη τη λισαβόνα έχει αποτύχει παταγωγό, τιμάζετε την ευρωπαϊκή επιτροπή 2020 ω διεύρυνση ω συνέχεια αυτή τη συνθήκη. αντιμετωπίζετε κύριε πρόεδρε την Ελλάδα ω τον αποδιοπομπαίο τράγο, υπαγορεύοντα μέτρα κατά των εργαζόμενων που δεν φταίνε για την κρίση, που όμω αυτά τα μέτρα θα είναι προπομπό για μέτρα και για τι άλλε χώρε. Ο λαό τη Ελλάδα και οι ευρωπαϊκοί λαοί σε λίγο καιρό θα σα αντιμετωπίζουν όπω αντιμετώπισε ο, ο λαό τη Αργεντινή στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι συμβολικό ότι 20 χρόνια μετά την κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσματος στην Ευρώπη μιλούμε για την Ευρώπη του 2020. Έχουμε δύο 20 δηλαδή, χρόνια μετά το τέρμα του διχασμού. Μιλούμε για καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, αηφόρο, οικονομία. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ την ανάπτυξη των υποδομών και μια αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική. Νομίζω ότι η σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και η διαφοροποίηση της ενεργειακής προμήθειας, του ενεργειακού εφοδιασμού. Ας μην ξεχνούμε σημαντικά σχέδια όπως ε, το Via Baltica και το Rail Baltica, που είναι σημαντικά όχι μόνο για τη Λιθουανία. Χρειαζόμαστε στη νέα στρατηγική μας ε, να αξιολογήσουμε τους λόγους ε, για τους οποίους δεν υλοποιήσαμε τους προηγούμενους στόχους της Λισαβόνας. Χρειαζόμαστε ρεαλιστικούς στόχους για την επόμενη στρατηγική, αλλά και να περάσουμε από τα λόγια στα έργα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σώσα Βάγνερ. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η κρίση αυτή νομίζω ότι μας δίνει μια ευκαιρία για να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα και πεποίθηση προκειμένου να διαμορφώσουμε μια ισχυρή Ευρώπη. Σε αυτή την ισχυρή Ευρώπη πολύ πιθανόν ε, να μην χρησιμοποιούμε τον όρο βελτίωση του συντονισμού. Γιατί Πολλέ φορές με το πρόσχημα του συντονισμού οδηγούμαστε σε ακινησία και παράλυση. Γνωρίζουμε ότι τα οικονομικά και τα δημόσια χρέη των χωρών μελών θα υποφέρουν αν δεν βαδίσουμε προς ε, μια δημοσιονομική ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και δεν ε, εκδοθούν ευρωομόλογα. Νομίζω ότι τα κοινοτικά θεσμικά όργανα μπορούν να προβούν σε συγκεκριμένες δράσεις και να μην θεωρητικολογούν με τον συντονισμό. λάβει το στην κυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριε Κύριε Λάγεν, καθίστε, σταθείτε μάλλον μπροστά στο μικρόφωνο στην θέση στο έντρανο υπαριθμό 40 και θα σας ανοίξει το μικρόφωνο ο τεχνικός. Wer würde das wagen, Herr Langen? Das... Gehen Sie bitte zu... Στην θέση σας, στο 40 παρακαλώ, Επιστρέψτε και ο τεχνικός θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα. Υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, όπως ε, καταλάβατε όλοι. Θα περιμένουμε λίγο. Ο κύριος Λάγκεν μπορεί να κάνει λίγο εξάσκηση, να σταθεί μπροστά στο μικρόφωνο. Όχι, να μην τραγουδήσετε αν θέλετε. Δεν μην τραγουδήσετε. Θα σας τα αφαιρέσουμε από το χρόνο μιλία Να ξαναδοκιμάσουμε. Ο τεχνικός προσπαθεί να το λύσει το πρόβλημα. Γιατί να τώρα, δεν θα πούμε στη συζήτηση γιατί παρουσιάστηκε το πρόβλημα στον κύριο Λάγκη συγκεκριμένα. Το 40 ξαναπροσπαθήστε. Nochmal bitte. bitte. Α, εδώ μάλιστα, εδώ μάλιστα. Δεν ξέρω αν λύθηκε και το πρόβλημα τη διερμηνία, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τεχνική λύση. Αν η στρατηγική της, αν η στρατηγική της Λισαβόνας για το 2020 θέλουμε να πετύχει, μάλλον αν η στρατηγική για το 2020 θέλουμε να πετύχει, θα πρέπει να διαμορφωθεί διαφορετικά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν ήταν η στοχοθέτηση λάθος. Τα κράτη-μέλη απλά δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους, τους κανόνες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε δεν επέτυξε το απαραίτητο θάρρο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, στην εφαρμογή της στρατηγικής της και με μεγάλη πλέον πλειοψηφία εξελέγει η δεύτερη επιτροπή. Ελπίζω να βελτιωθούν όλα αυτά, να υπάρχει πιο πολύ δυναμισμό στην Ευρώπη, να μην μιλάμε για ανακατανομή μόνο, αλλά να είναι καλύτερη η ανταγωνιστική μας θέση στον κόσμο. η δική μας απάντηση ε, θα πρέπει να είναι δυναμική. Αυτό θα πρέπει να περιέχει η στρατηγική αυτή. Και θα πρέπει να πω ότι ως τώρα έχω δει μόνο σχέδια γιατί... και ελπίζω να βελτιωθεί αυτό το σχέδιο γιατί αυτά που έχω δει ως τώρα αποτελούν μια συνέχεια της προηγούμενης κατάστασης και δεν άκουσα και κάτι καινούργιο ιδιαίτερα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, αλλά χρειαζόμαστε τη στρατηγική αυτή για να αντέξουμε και θα πρέπει να οριστούν νέοι όροι, θα πρέπει να συζητηθούν οι κλιματολογικοί όροι του παρελθόντος, θα πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συνολικό όργανο να μην εκπροσωπεί μόνο τα συμφέροντα των ε, επιτρόπων, αλλά να αναλάβει την ηγεσία στην Ευρώπη. Για να είσαστε βέβαιοι, αν συμβεί αυτό, θα έχετε την αμέριστη και την ανεφόρον ε, ε, υποστήριξή μας. Όχι όμως να συνεχιστεί αυτή η ατολμία των κυβερνήσεων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λεφόλ. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε Βαρόζο, κύριε Πρόεδρε Βαν Ρόμποϊ, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι για την στρατηγική του 2020 όλοι συμφωνούμε ως προς τους στόχους. Το πρόβλημα όμως στην Ήπειρο μας σήμερα είναι ότι ε, ξέρχεται από μια σοβαρότατη κρίση που το χαρακτηριστικό της είναι μια αδύναμη για να μην πω αρνητική ανάπτυξη. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια πολιτική συνειδητοποίηση της κατάστασης με δύο στόχους. Καταρχήν, πώς θα διοργανωθούμε πολιτικά για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Στα δικά σας αξιώματα θα πρέπει να υπομειστείτε δύο ευθύνες. Καταρχήν, να προβείτε σε ένα συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, να καθορίσετε στόχους με συγκεκριμένα εργαλεία για την υλοποίησή τους. Και έρχομαι εδώ στο δεύτερο σημαντικό κατά τη γνώμη μου σκέλος, που έχει τη μορφή ερώτησης για να, υλοποιηθεί, υλοποιηθούν στόχοι σε μια δημόσια πολιτική χρειάζεται προπολογισμό. Και αυτό το δίλημα έχουμε σήμερα. Οι χώρε έχουν πολύ σημαντικά ελλείμματα και όσο σημαντικότερα είναι τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τόσο λιγότερα θέλουν να προσφέρουν στον κοινοτικό κοροβανά. Γι' αυτό με ισχνού προπολογισμού πώ θα προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη, Πώ θα λύσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό, αυτό το δίλημα. Ποιε είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ, που θα υποστηρίξετε στη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές απέναντι στα κράτη-μέλη. Έχετε τη δυνατότητα, την ικανότητα να προτείνετε καινοτομίες ώστε και η Μπερτ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να λάβουν περισσότερες ευθύνες και να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δανειστεί για να χρηματοδοτήσει την ανάγκη αυτή, να υλοποιήσει την οικονομική της ανάπτυξη. Η κυρία Γκουλάχ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. κύριε Πρόεδρε, μετά από τη στρατηγική της η ειδού η στρατηγική 2020 και είναι απλή αλλαγή ονομασία και λιγότερο αλλαγή κατεύθυνση. Και στρέφομαι κυρίω προ τον κύριο Μπαρόσο, διαβάζοντα τη συνεισφορά σα εν ώψη του τύπου συμβουλίου, ακούγοντά σα σήμερα να αναφέρεστε και σωστά στον αριθμό των φτωχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη να αναπτυχθεί ο χρηματοπιστωτικό κανονισμό. Σα λέω, κύριε Βαρόσο, κρίμα που δεν είσαστε πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια, διότι θα μπορούσατε να κάνετε όλα αυτά που μα προτείνετε σήμερα και σήμερα μα λέτε ότι είναι η κρίση που σα εμπόδισε να τα κάνετε, αλλά η κρίση λοιπόν σε κάτι οφείλεται. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να χάνουμε τώρα τον χρόνο με δηλώσει ευλαχνία. Τώρα προ τον κύριο Βανρομπόη, καταρχά να, ευχα... να του πω με πιο ευγενικό τρόπο το απλώ ήρθε σε σχέση με αυτά που άκουσα από κάποιου βουλευτέ, από ένα βουλευτή προηγουμένω. Σε εσά βασιζόμαστε. Είναι παράδοξο, κύριε Βαρομπόη. Θα ε, βασιζόμαστε σε μια πραγματική κοινοτική Ευρώπη να πορευθούμε και ξέρουν οι χώρες, η χώρα μου ξέρει τι σημαίνει κοινοτική Ευρώπη. Λοιπόν, εάν κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση θα έχετε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου μα και η στρατηγική του 2020 δεν θα πρέπει ε, να παραμείνει απλώ λέξει. Αν έχουν νόημα οι λέξει, θα πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται μεσοπρόθεσμα σε σφαιρικό επίπεδο πέρα από του εθνικισμού. Συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Λάμπερτ. Τα μέλη του Συμβουλίου για την χρηματοστηρική εποπτεία δεν μα δίνουν αυτή τη στιγμή μεγάλα ευρωπαϊκά οράματα και βάζουν και τα δύο πόδια στο φρένο. Λοιπόν, θα ήθελα να πετύχουμε αυτά που είπατε και στο έγγραφό σα στο Συμβούλιο. Θέλουμε μια οικονομική και νομισματική Ευρώπη με όλε τι πτυχέ Να ε, υπάρχει πειθαρχία, αλληλεγγύη, να παγιωθούν επενθυμιστεί στο Συμβούλιο ότι αν υπάρχουν προβλήματα στην Ελλάδα, εν μέρη οφείλονται στου Έλληνε και εν μέρη στην έλλειψη αλληλεγγύη οφείλονται. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σμπουτικόφερ. Ένα μισή λεπτό. Είναι εύκολο να θέτουμε ωραίους στόχους. Όλοι μας θέτουμε ωραίους στόχους στην αρχή του κάθε χρόνου, αλλά το να είμαστε πιστοί ε, στους στόχους και το αν ε, θα εξελιχθούν αυτοί σε πραγματική ατζέντα εξαρτάται από το ποιος, πότε, πόσο, πότε θα γίνουν όλα αυτά. Και όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε, θα φανούν σε ό,τι αφορά την στρατηγική για το 2020. Στην αρχή της συζήτησης ο κύριος Ντόιλ νομίζω ότι έθιξε το πιο σημαντικό θέμα. Το πιο σημαντικό θέμα είναι κατά πόσο είμαστε διτεθειμένοι να εκχωρήσουμε στο θέμα της οικονομικής πολιτικής την εθνική αρμοδιότητα ή προτιμούμε να εκχωρήσουμε συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ζώνη του ευρώ, να εκχωρήσουμε αυτά που έχουμε πετύχει τόσες δεκαετίες. Αυτό είναι το δραματικό, εναλλακτικό σενάριο. Μου έκανε εντύπωση που άκουσα από τους χριστιανοδημοκράτες τόσο σαφή λόγια γιατί είναι οι συντηρητικοί στη Γερμανία αυτοί οι οποίοι ανακόπτουν την πορεία αυτή εδώ και καιρό στην ε, Γερμανία. Θα ήθελα να πω το εξή. Ελπίζω να μην είναι μόνο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που βγαίνει και λέει ότι θέλει το Συμβούλιο να δώσει κατευθυντήριες οδηγία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Κοινοβούλιο να δραστηριοποιηθούν ενεργά προς την κατεύθυνση αυτή, προς την κατεύθυνση μιας κοινή ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, η οποία δεν θα είναι μόνο, αν θέλετε, εμπορική συμφωνία Σαρκοζή Μέρκελ, αλλά θα είναι μια σοβαρή προσπάθεια κοινή διακυβέρνηση της Ευρώπης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο κύριος Αγκουράκης. Ένα λεπτό. Ε, την ώρα που εμείς ε, συζητάμε κυρία Πρόεδρε τα αποτελέσματα της έκτακτης συνόδου κορυφής όπως γνωρίζετε πολύ καλά στην Ελλάδα όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς εξαίρεση απεργούν καταγγέλλοντας ακριβώς αυτά τα μέτρα αυτά τα αποτελέσματα καταγγέλνουν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική των κεντροαριστερών και κεντροδεξιών κυβερνήσεων που ομοφωνούν στην λήψη αντιλαϊκών αντιεργατικών μέτρων για να διασφαλίσουν αποκλειστικά και μόνον τα κέρδη των μονοπωλίων. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσει και επιτροπή προσπαθούν να τρομοκρατήσουν του εργαζόμενου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποκύψουν στην αντιλαϊκή θύελα. Στον πόλεμο αυτό οι εργαζόμενοι απαντούν όμω με μαζικέ απεργίε, διαδηλώσει και κινητοποιήσει για τι οποίε δεν άκουσα τίποτα να λέτε κύριε Μπαρόσο, με, ε, διαδηλώσει και απεργίε που οργανώνουν τα ταξικά συνδικάτα σε πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μέτωπο των κομμάτων του κεφαλαίου του ευρωμονόδρομου των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών στη γενικευμένη επίθεση της κυβέρνησης στους μισθούς και συντάξεις μία μπορεί να είναι η απάντηση των εργαζομένων μία ανάπτυξη ε, προς όφελος των δικών τους συμφερόντων. Ο κύριος Μπορκέζιο, ένα λεπτό. Λοιπόν, ε, εκφράζουμε επίσημα αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, αλλά τελικά εφαρμόζεται μια πολιτική αυστηρότητα στην πράξη όσον αφορά τα κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Βαν Ρομπουή στην συνέντευξη τύπου είπε σαφώ ότι η ιδέα είναι να σταθεροποιηθεί ένα είδο δικτατορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μετατρέποντα να γίνει χούντα το Συμβούλιο με μεγαλύτερε εξουσίε εναντί των κρατών μέλων. Πριν από τη Σύνοδο Κορυφή, αποκάλυψε η Independent, έστειλε μια επιστολή στου αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων και έλεγε σε κάποια από του παραγράφου τα μέλη του Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τι οικονομικέ στρατηγικέ των κυβερνήσεών του, πρέπει να κάνουν το ίδιο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και ζητά συντονισμό τη οικονομική πολιτική μόνο στο Συμβούλιο, ούτω ώστε να διαμορφώνεται και να υποστηρίζεται μια στρατηγική ευρωπαϊκή εκεί. Και προσθέτει το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό είναι πολύ φιλόδοξο. Θέλουμε να είμαστε, κυρία Χιν, να προσανατολίζουμε, να κατευθύνουμε και γι' αυτό εγώ πρότεινα να συνεδριάζει κάθε μήνα το Συμβούλιο. Έχει αυτοκρατορικέ προσδοκίε, τελικά το Συμβούλιο και εκφράζεται μέσω μια ε, μιας προτάσεως που κυκλοφορεί στους διαδρόμου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζητεί το 80% του χρέου των μελών, 100 μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσης να γίνει χρέο τη Ευρωπαϊκή Ένωση η εκστρατεία για μια επικυβέρνηση οικονομική που προγραμματίζεται αυτές τις μέρες κινδυνεύει να μεταμορφώσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε προτεκτοράτα. 1,5 ε, λεπτό, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε λοιπόν μια στρατηγική μετά τη Λισαβόνα, χωρίς να έχει θέσει όμως ε, ε, μετρήσιμους στόχους. Μόνο και μόνο για να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χρειαζόμαστε καλά εξειδικευμένες δυνάμεις ε, και όχι διαδοχικά μεταναστευτικά ρεύματα τα οποία πλημμυρίζουν τις εθνικές αγορές και αν θέλουμε πιο ευέλικτη διαμόρφωση των εθνικών αγορών αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση των προθεσμιών σε ό,τι αφορά τα νέα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης όπου απειλείται η δουλειά πολλού κόσμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εγκαταλείψει τα μέτρα ανταγωνιστικότητας. Και γενικά δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυθαιρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χρειαζόμαστε δεν χρειαζόμαστε σε καμία περίπτωση νέες εξετάσεις, νέα έγγραφα για τους στόχους αυτούς που θα καταλήξουν σε συρτάρια. Χρειαζόμαστε επιστροφή σε εθνικές αρμοδιότητες. Δεν μπορεί το, η Ευρώπη του 2020 και η σχετική στρατηγική παρά να εξυπηρετήσει τον Ευρωπαίο πολίτη. Θα πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιαστεί όσο χειρό κατά της παγκοσμιοποίησης. Ο κύριος Μάουρο λέει πρόεδρος για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, ίσως δεν θα είσαστε πολύ γνωστός όπως υποστηρίζει ο κύριος Φάρατζ. Αλλά ξέρω ότι τα ιδεώδη σας ε, ριζώνονται στις παραδόσεις της Ευρώπης, στον πολιτισμό της Ευρώπης και στη... σας εκτιμώ γι' αυτό και σας σέβομαι. Επιτρέψτε μου όμως να σχολιάσω την παρέμβασή σας που ήταν πάρα πολύ ορθολογική συγκρίνοντάς το με τον ποδόσφαιρο. Αυτά που είπατε. Το όραμα που έχετε εσείς όσον αφορά το ρόλο σας θεωρώ ότι είναι παρόμοιο με ενός παίκτη του κέντρου, του κέντρου που είναι μέτριο στο παιχνίδι της ομάδας και μετά την αλλαγή των κανόνων που επιβάλλει η συνθήκη της Σαββόνας μπορεί να είναι πιο δύσκολο να πετύχει τέρμα, να πετύχει τους στόχους τους γιατί αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Υπό το φως αυτού του παραδείγματος πιστεύω ότι στο κοινοβούλιο να απόκειται να κινδυνεύει περισσότερο από τους άλλους παίκτες. Να είναι κάποιος που έχει φαντασία εφάνταστος παίκτης που εφευρίσκει το παιχνίδι βασιζόμενο στους νέους κανόνες για να αυξήσει την επιθετική δυνατότητα της ομάδας και ο, αυτός ο κεντρικός παίκτης μας που είναι επιτροπή του κυρίου Μπαρόσο να είναι σε θέση τελικά να σκοράρει. Ε, τι θα συμβεί αν δεν ακολουθήσουμε αυτή την τοποθέτηση που εγώ συμμερίζομαι σε μεγάλο βάθος. Θα κλειστούμε στην άμυνα στο παιχνίδι και θα σημειώσουμε αυτόν γκολ ε, εναντίον των συμπολιτών μας. Λοιπόν, γι' αυτό σας ζητώ κύριε Πρόεδρε να υποστηρίξετε το νέο πρωταγωνιστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μην το βλέπετε αυτό σαν εμπόδιο, αλλά σαν μια ευκαιρία, μια δυνατότητα. Είμαστε όλοι μαζί που καλούμαστε σε ιστορικές περιστάσεις να διαδραματίσουμε ιστορικό ρόλο, ιστορική αρμοδιότητα. Είμαι σίγουρος ότι είσαστε ο σωστός άντρας για να μας κατευθύνετε. Σας ευχαριστώ κύριο Λόπες Αγγιλάρη για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, μιλούμε για τη στρατηγική του 2020 ουσιαστικά για όχι μόνο για τη στρατηγική μετά τη Λισαβόνα, αλλά για τη στρατηγική της αναγνώρισης της α, ε, αποτυχίας της Λισαβόνας, για να το πούμε ομά και ειλικρινά. Γιατί κανονικά η Λισαβόνα έπρεπε να εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την αηφορία. Δεν τα κατάφερε όμω. Ούτε αηφορία εξασφάλισε οικονομική, δημοσιονομική, ούτε κοινωνική, ούτε περιβαλλοντική αηφορία. Από οικονομική και χρηματοοικονομική άποψη κατασκευάσαμε την νομισματική Ένωση, αλλά ούτε καν συντονισμό τη οικονομική πολιτική και των φορολογικών κινήτρων που πρέπει να συνοδεύουν μια νομισματική πολιτική δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε. Από ενεργειακή άποψη, η ενότητα τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι ανύπαρκτο. Και από κοινωνική άποψη, δυστυχώ, ε, ε, είναι αισθητή στην Ευρώπη. Η δυσαρέσκεια των εργατών, των συνδικάτων και των πιο μειονεκτικών στρωμάτων τη κοινωνία που ανησυχούν για το κατά πόσο είναι βιώσιμο αυτό το μοντέλο που εξασφάλιζε κάποια στιγμή ευημερία και κράτος πρόνοιας και μας χαρακτήριζε ως Ευρωπαίους. Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου τι δέσμευση θα αναλάβει μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχυθεί αυτή η δέσμευση με το προς το κοινωνικό μοντέλο ένα θέμα που είναι προσφυλές στην ασκούσα την Προεδρία Ισπανική Προεδρία, όπως μας είπε και ο Χωσέ Θαπατέρο. Θέλουμε ένα κοινωνικό μοντέλο που να λέει ότι η Ευρώπη είναι υπέρ της περιβαλλοντικής, δημοσιονομικής σταθερότητας και της προάσπισης ε, της ε, κοινωνικής ευημερίας και του κοινωνικού ευρωπαϊκού μοντέλου που μας χαρακτήριζε. Ο κύριος Λάμπερτ, ένα λεπτό. Ο κύριος Παρόσο είπε, μίλησε προηγουμένω και είπε ότι θέλει μια φιλόδοξη στρατηγική. Αληθεύει ότι υπάρχουν κάποια τμήματα τα οποία της στρατηγικής του 2020 που είναι φιλόδοξα, αλλά σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών δεν μιλάμε για φιλοδοξού στόχους. Δεν θα μας οδηγήσουν αυτά τα νούμερα στους ε, στόχους που θέλουμε. Θα πρέπει να περικόψουμε κατά 40% μέχρι το 2020 και μιλώντα για το κλίμα θα πρέπει να δούμε και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. Επίσης πολλά φαίνεται να επαναλαμβάνονται στη στρατηγική αυτή σε ό,τι αφορά οικονομική, την οικονομική ανάπτυξη, η οποία α, τίθεται ως στόχος, όχι ως ένδειξη, όχι ως δείκτης. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλούς τομείς όπου προσπαθούμε να αποσυνδέσουμε την ανάπτυξη από τη μεταφορά για παράδειγμα και αυτό έχει αποσυνδεθεί από τις θέσεις εργασίας. Άρα σας παρακαλώ μην μας λέτε ότι η ανάπτυξη θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Το θέμα δεν είναι να μειώσουμε μόνο τη φτώχεια αλλά και τις ανισότητες γιατί αυτό θα έχει σκοπό. Θα πρέπει να μην υποσκάπτουμε τους φιλοδοξούς στόχους που μπορεί να επιβάλλουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καράς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Θα ήθελα καταρχάς να σας ε, ευχαριστήσω για την επιστολή που μας αποστήλατε. Θα ήθελα να σας πω ότι Συμφωνώ με τις αρχές που αναφέρετε 100% της προσυπογράφω. Χαίρομαι που είπατε ότι θέλετε να συνεδριάζετε σε μηνιαία βάση, γιατί σκοπό σας και καθήκον σας είναι να πλησιάσει ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπήρξε έλλειψη πολιτικής βούλησης για την εφαρμογή των στόχων αυτών σε κάθε χώρα. Εσάς δικό σας καθήκον θα είναι ο συντονισμός των κρατών μελών στο σημείο εκείνο όπου υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής, μάλλον που δεν αρκεί η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπατε σαφώς ότι δεν αρκεί ε, η αγορά. Θέλουμε κοινωνική ε, ε, οικονομία της αγοράς, αλλά χρειαζόμαστε και πολιτική ένωση. Και το πρώτο, η πρώτη πρόκληση θα είναι ο προϋπολογισμός του 2011. Και θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτό η στρατηγική του 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 δεν αποτελεί αυτό σκοπό, αποτελεί το μέσο για να πετύχουμε όλα εκείνα τα οποία θέλουμε να δώσουμε ως απάντηση στην χρηματοοικονομική κρίση. Ναι, χρειαζόμαστε πιο πολύ συντονισμό με την δημοσιονομική, στη δημοσιονομική, στη φορολογική πολιτική, στην πολιτική για την εκπαίδευση, για την έρευνα, την ανάπτυξη. Γιατί δεν ε, επιτυχάνεται μόνο η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα με οικονομικούς στόχους και χρειάζεται και εφαρμογή του Small Business Act ε, στα κράτη-μέλη. Small Business First, γιατί έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας ε, στις περιφέρειες και θα ήθελα να σας καλέσω να ζητήσετε μία μελέτη αντικτύπου για να δείτε Ποιο ήταν ο αντίκτυπο όχι μόνο στι τράπεζε, αλλά και στην κοινωνία. Να δούμε ποιε ε, είναι οι εξελίξει που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τι συντάξει ε, για, τον πληθυσμό και το καθεξής. Και όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στα πλαίσια του 2020. Ευχαριστώ κύριε Κάρας, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Σέρκας, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμένα μου άρεσε πολύ η μελωδία που ακούσαμε σήμερα. Ελπίζω και η στίχη του τραγουδιού την επόμενη εβδομάδα να είναι αντάξει της μελωδίας. Αυτό θα σημαίνει ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί και εσείς και εμείς ότι δυνάμεθα και οφείλουμε να καθορίσουμε κάποιους στόχους και μπορούμε να επιλέξουμε το μέλλον μας. Δεν υπάρχει κανένας οικονομικός δετερμινισμός. Υπάρχει μία φωνή για την πολιτική, υπάρχει μία φωνή για τους πολίτες, για το μέλλον μας και το μέλλον βρίσκεται στα χέρια μας. Η οικονομία μας δείχνει κάποια όρια σίγουρα, αλλά μας δίνει και κάποια μέσα ταυτόχρονα. Οι στόχοι είμαστε εμείς οι ίδιοι και θα πρέπει ε, η οικονομία να εξυπηρετεί την κοινωνία και όχι το αντίστροφο. Όπως ακούσαμε σήμερα το απόγευμα, χρειαζόμαστε μια μακρόπνοη, μακροπρόθεσμη στρατηγική και όχι μόνο μια κοντόφθελμη και βραχυπρόθεσμη στρατηγική. Αυτό ήταν το δίδαγμα του παρελθόντος. Είχαμε πολύ σημαντικά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης στο παρελθόν, αλλά με κερδοσκοπικές βάσεις που δεν έλαβαν υπόψη τη δικαιοσύνη, την ισότητα, το περιβάλλον, το μέλλον των επερχόμενων γενεών. Μακάρι κύριε Πρόεδρε την επόμενη εβδομάδα να υποβληθούν έγγραφα με φιλόδοξο πρόγραμμα που θα δίνει έμφαση στην αηφορία που θα εξασφαλίσει τη συμφιλίωση του οικονομικού, του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού σκέλους, γιατί υπάρχει συμβατότητα μεταξύ τους. Επίσης, προσοχή στην κοινωνική διάσταση του προγράμματος, γιατί εκεί αποκρισταλώνονται οι αιτήσει, οι αξιώσεις, ε, τα όνειρα και οι προσδοκίες, αλλά και οι φόβοι των Ευρωπαίων πολιτών. Οι φόβοι αυτών που έμειναν εκτός της ε, ε, αγοράς εργασίας, τα θύματα της αλαζονίας των χρηματοπιστωτικών αγορών προσβλέπουν σε, στην σε εμά για να βάλουμε κάποια όρια, για να κάνουμε ποιοτικέ θέσει απασχόληση προσιτέ σε όλου, ώστε ε, χαρακτηριστικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η αριστεία και όχι η πάλι για την ε, συρρήκνωση των κοινωνικών προδιαγραφών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίγκολ, ένα λεπτό. Αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμη πρόεδροι. Καταρχάς, η κρίση της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας είναι τόσο βαθιά που στην κατάσταση αυτή πραγματικά περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Συγκεκριμένες προτάσεις α, προς την κατεύθυνση που διατυπώθηκαν, που από πολλούς ε, βουλευτές. Περιμένουμε μία πρόταση για το πώς ε, οι κίνδυνοι υψηλής χρέωσης ε, μπορούν να αποφευχθούν προκειμένου η Ελλάδα και άλλοι να μην καταπιεστούν υποβάλλετε προτάσεις όπως ε, ζήτησε χθε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το πώς θα μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και δεν θα πρέπει να τιμωρούνται μόνο οι χώρες με έλλειμμα αλλά και οι χώρες με επιβολικό πλεόνασμα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία τα οποία θα είναι ανεξάρτητα και θα είναι ανεξάρτητα και από τις φορολογικές πολιτικές έχει κάνει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η σειρά σας πλέον να θέσετε συγκεκριμένες προτάσεις. Ο κύριος Οντί, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτέλους σας είδαμε κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Καλώς ήρθατε στην Ολομέλεια. Πάντως ε, αισθάνομαι ε, τεράστια απογοήτευση που δεν ήταν ε, το πρώτο σας διάβημα να έρθετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την 1η Δεκεμβρίου μόλις τώρα σας βλέπουμε στην Ολομέλεια. Κρίμα. Εδώ ασκούμε πολιτική και πολιτική χωρίς δημοκρατία δεν νοείται. Γιατί μην ξεχνούμε τα γαλλικά και ολλανδικά δημοψηφίσματα, αλλά και άλλα δημοψηφίσματα να γίνονταν, θα ακούγαμε από τους Ευρωπαίους πολίτες όχι ότι είμαστε κατά της Ευρώπης, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι η Ευρώπη γίνεται ερήμην μας και μερικές φορές εις βάρος μας. Ευχαριστώ. Βέβαια, η Άγγελα Μέρκελ και ο Νικολάς Σαρκοζή έφεραν ευτυχώ τον πολίτη στο επίκεντρο και στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, που δημιούργησε και το αξίωμα που καταλάβατε εσεί, κύριε Πρόεδρε. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρί του πολίτε και χωρί του εκπροσώπου των Ευρωπαίων πολιτών. Επίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αντιληφθεί ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρί τα κράτη και του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Α έρθουμε όμω στο ψαχνό. Οι Ευρωπαίοι πολίτε υποφέρουν γιατί δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το νόημα τη παγκόσμια ταραχή. Θα πρέπει να τους δώσουμε ένα μπούσουλα, μια κατεύθυνση για να δουν ότι η Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημα, είναι η λύση, ότι δεν τους εκθέτει, τους προστατεύει, δεν την υφίστανται, αλλά τους δίνει περιθώριο λιγμών. Ποια είναι η θέση τους στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ποιο τμήμα, τι τμήμα θα δώσετε στο διακυβερνητικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση που αυτή τη στιγμή λείπει και στην σύσταση και ίδρυση της εξωτερικής υπηρεσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο πόδια, τα κράτη και τις κυβερνήσεις αφενός και τους πολίτες αφετέρου. Εσείς είστε το κεφάλι, δεν θα πρέπει να είστε στην δεύτερη θέση, αλλά στην πρώτη θέση. Εσείς θα πρέπει να διευκολύνετε την αλληλοβοήθεια μεταξύ των χωρών μελών σε μια πολιτική ένωση. Από αυτή θα εξαρτηθεί το μέλλον της Ένωσης. Σας ευχαριστούμε που είστε στη θέση σας. Έχετε πολλά προσόντα. Μη φοβάστε τους πολίτες και τους εκπροσώπους τους. Αλλά να ανοίξετε τους στην όλη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριο Σκοφεράτη. Για ένα μισή λεπτό, συγγνώμη κύριο Σκοφεράτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κατά τον καθορισμό της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020 θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης που αυτή τη στιγμή ταλανίζει αυτό το τμήμα της Ευρώπης και όχι μόνο. Και τα όρια που καθόρισαν τα μέτρια αποτελέσματα της στρατηγικής της Λισαβόνας του 2000 η κρίση μας δίνει σαφές ενδείξεις όσον αφορά την ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση αν θέλουμε να θέσουμε όπως θεωρώ αναγκαίο αυτό το στόχο εντός των δρασεών μας. Εν πρώτης, χρειάζονται μέσα ρυθμιστικά για υποπτία των χρηματοστικών συστημάτων των τραπεζών, ούτω ώστε να μην ξαναδημιουργηθούν οι συνθήκες οι αρνητικέ εκείνες που μας οδήγησαν σε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να έχουμε μεγάλες επενδύσεις διαθέσιμες για την έρευνα, την καινοτομία και την ε, ενημέρωση, αν θέλουμε να κατευθυνθούμε προ την ανοιχτή αγορά κυρίω. Αλλά αυτές οι μεγάλες επενδύσεις για να γίνουν η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ευρωομόλογα και ένα σύστημα ε, ε, κυρώσεων για την επίτευξη των ε, και κινήτρων για την επίτευξη των οικονομικών στόχων. αυτή πρέπει να είναι οι στόχοι που έλειπαν και χρειάζεται να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή όσον αφορά τα έσοδα, όσον αφορά του μισθού και την φορολόγηση. Χρειάζεται συντονισμένη βιομηχανική πολιτική κατά τομέα για να υπερασπιστούμε την παραγωγική δομή, την κατασκευαστική που είναι ιστορική αξία ε, στην περιοχή μα. Και τέλο, θα πρέπει να ξαναδιαμορφωθεί ο κοινωνικό διάλογο σαν ένα στοιχείο συνοχή και συγκράτηση των κινδύνων από την ανεργία μακρά διαρκείας, κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Καλούμε θα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Τηλικαστή δύο λεπτά. Eh, <clears throat> eh, Σα ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε Ρόμπε, κύριε Πρόεδρε Μπαρόζο, απουσιάζει βέβαια. Θα ήθελα να αποταθώ όμω και σε εκείνον. Χαίρομαι που ήρθατε και οι δύο μαζί πολύ ευχάριστη αυτή η εικόνα και χαίρομαι που υπάρχει μια προσέγγιση και μια προσήλωση στα θεμέλια, μια κοινή προσήλωση στα θεμέλια της μελλοντικής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη του 2020. Αυτό που περισσότερο τράβηξε την προσοχή μου και το ενδιαφέρον μου από τη γραπτή σας πρόταση είναι ότι οι στόχοι θα πρέπει να είναι λίγοι, να περιοριστούμε στις προτεραιότητες, να είναι χειροπιαστή η στόχη αυτή, να μπορούν να αποσυντοκοπηθούν, να αξιολογηθούν και να καταμετρηθούν συστηματικά για να δούμε κατά πόσο σημειώνουμε πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι σημαντικό να γίνεται αυτή η τακτική αξιολόγηση και συνιστά μια ποιοτική αλλαγή ουσιαστική σε σχέση με την προηγούμενη στρατηγική της Λισαβόνας. Εγώ θα επιμείνω σε ένα στόχο, την εσωτερική αγορά Πάνε πάνω από 20 χρόνια που η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ε, σχεδιάστηκε και άρχισε να εφαρμόζεται. Έχουν περάσει όμως 20 χρόνια και δεν έχουμε υλοποιήσει μια πραγματικά εσωτερική αγορά στους περισσότερους τομείς. Σε ορισμένους κλάδους βέβαια, όπως είναι ο ψηφιακός, ε, οι εμπειρίες μας είναι πολύ πρόσφατες. Αλλά ακόμη και σε άλλους τομείς έχουμε τέτοιο κατακαιρματισμό, τόσους φραγμούς και εμπόδια, που στερούμε από την ευρωπαϊκή οικονομία το μέγεθος κλίμακος που χρειάζεται για να, για να μπορέσει πραγματικά να αναπτυχθεί, να γίνει ανταγωνιστική και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη. κύριε Βαρόμπεο και Μπαρόζο, χρειάζεται σημαντική πολιτική όθηση. Το σαν να μην συνέβη τίποτα, το business as usual δεν αρκεί πια. Χρειάζεται ηγετικός ρόλος και φυσικά ανάληψη ευθύνη. Μπορείτε να υπολογίσετε στην αμέριστη υποστήριξή μου για να το υλοποιήσετε. Ευχαριστώ κύριε Μπούλμαν. Ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δύο σημεία θα ήθελα να θίξω, πολύ συγκεκριμένα. Καταρχάς, έχουμε ήδη μία φιλόδοξη στρατηγική που θα υπόσχεται την ε, επιτυχία σε ό,τι αφορά το 2020. Όχι. Και να σας πω γιατί. Γιατί αν λέτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν λέμε στα κράτη-μέλη ότι πρώτα θα κάνουμε την ενίσχυση του προϋπολογισμού και μετά θα κοιτάξουμε την οικονομία και την απασχόληση, πρόκειται πολύ απλά για μια εξίσωση η οποία δεν βγαίνει. Αν δεν μας πιστεύετε, διαβάστε τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην τοποθέτησή του χτες. Ότι υπάρχει ανησυχία για τη διεθνή κατάσταση. Αν δεν τεθούν ε, λοιπόν συγκεκριμένοι στόχοι απασχόληση, δεν θα αντιμετωπίσουμε ποτέ την κρίση. Κατά δεύτερον, έχουμε απάντηση σε ό,τι αφορά την κρίση του, της υπερχρέωσης των χωρών που έχουν πληχθεί. Όχι, όχι, δεν έχει δοθεί απάντηση. Άνα, αν διαβάσετε τα στοιχεία της ανάλυσης, θα καταλάβετε ότι τουλάχιστον ε, τα μισά οι μισές υπερβολικές δαπάνες της Ελλάδας οφείλονται σε κερδοσκόπους. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, το οποίο θα συνδράμει τις χώρες αυτές, οι οποίες έχουν ανάγκη. Δεν χρειάζονται μόνο βοήθεια χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαζόμαστε μάλιστα τη βοήθεια αυτή εδώ και τώρα, κύριε Μπούλμαν. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέρι, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, σαν μέλος της, του Προεδρικού Τρίου, σαν ε, ουγγρικό ε, μέλος της Βουλής θέλω να ευχηθώ στο νέο πρόεδρο του Συμβουλίου να κινηθεί προς τους στόχους της Ευρώπης. Είναι ένα σταυροδρόμι τώρα αυτό που βρισκόμαστε. Εκεί θα δούμε πώς θα λειτουργήσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αντιμετωπίζει κρίση η Ευρώπη και χρειάζεται σταθερό χέρι και κατεύθυνση. Είναι θέμα αξιοπιστίας αυτό που τίθεται. Το νέο πρόγραμμα που θα ακολουθήσει την ε, στρατηγική τη Λισαβόνα θα πετύχει. Εγώ κατάγομαι πρώην κομμουνιστική χώρα και εκεί σε αυτέ τι περιοχέ τη Ευρώπη υπάρχουν ε, κάποιοι δισταγμοί όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα ε, σχέδια. Δικαιολογημένο. Τώρα να αναφερθώ στη θεσμική διάσταση. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια θα είναι η νέα στρατηγική, ποιο είναι ο στόχο τη νέα στρατηγική, προ ποιου απευθύνεται η νέα στρατηγική. Αν θεωρούμε ότι απευθύνεται η στρατηγική στου πολίτε τη Ευρώπη που θέλουμε να του κερδίσουμε, και μαζί με τους οποίους θέλουμε να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική, πιο ισχυρή, αν αυτό θέλουμε, θα πρέπει να προχωρήσουμε σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα τη συνθήκη τη και θα πρέπει να συμμετάσχει πλήρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η σημερινή συζήτηση δεν αντικαθιστά την αντιμετώπιση και συζήτηση του θέματο και το να ακολουθήσουμε τι κανονικέ διαδικασίε, να υπάρξει κάποιο συζητητή και να διεξαχθούν συζητήσει στι επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την ουσία, στόχο θα πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων εργασία. Αυτή πρέπει να είναι αφετηρία κάθε νέα στρατηγική. Τώρα, πώ μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, είναι κάτι που δεν ξέρουμε πολύ καλά ακόμα. Ε, θα πρέπει να θεθούν προτεραιότητε, να υπάρξει στενότερο ίσω οικονομικό συντονισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα εξή. Καταρχά, αν θέλουμε θα πρέπει να βρούμε διορθωτικά μέτρα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να ισχυροποιηθεί λόγω κοινοτικών πολιτικών η Ευρώπη. Θα ήταν εσφαλμένο εάν κινηθούμε κατά των συνθήκων και να μην εφαρμόσουμε σωστή πολιτική συνοχή ή κοινή αγροτική πολιτική. Θα πρέπει όλε οι περιφέρειε τη Ευρώπη να ωφεληθούν στρατηγικέ και όχι απομονωμένε εταιρείε ή περιοχέ. Τρίτον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η στρατηγική αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα των κρατών μελών. Η κυρία Ποδηματά, δύο πραγματικοτητα των κρατων Δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έχουμε σήμερα εδώ για την στρατηγική του 2020, αλλά γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της 11 η Φεβρουαρίου κυριάρχησε το λεγόμενο ελληνικό ζήτημα. Και γνωρίζουμε επίσης ότι το έκτακτο αυτό Συμβούλιο Κορυφής κατέληξε σε μια δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων με την οποία παρέχεται πολιτική υποστήριξη στην ελλάδα εκφράζεται ετοιμότητα για ανάληψη δράσης για τη σταθερότητα του ευρώ και σημειώνεται ότι η ελλάδα δεν έχει ζητήσει οικονομική βοήθεια από την ευρωπαϊκή ένωση. και με την ευκαιρία θέλω να υπενθυμίσω ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο έλληνας πρωθυπουργός έχουν κατ' επανάληψη τονίσει ότι η ελλάδα δεν ζητάει χρήματα δεν ζητάει ούτε οι γερμανοί ούτε οι αυστριακοί ούτε οι σουηδοί ούτε κανένας άλλος ευρωπαίος φορολογούμενος να πληρώσει το χρέος της το οποίο θα το αντιμετωπίσει θα το περιορίσει στη βάση των δικών της προσπαθειών με βάση τα μέτρα που έχουν ήδη εξαγγελθεί και με την ευκαιρία αγαπητέ κύριε verhofstadt δεν είναι ακριβές ότι η ελλάδα έχει διαβεβαιώσει ότι έχει παράσχει όλα τα στοιχεία για το ομόλογο τη goldman ε, sachs έχει διαβεβαιώσει ότι θα τα παράσχει εγκαίρως αλλά με την ευκαιρία δεν βλέπω εδώ τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής πραγματικά θα ήθελα να εκφράσω την απορία μου γιατί ζητήθηκαν μόνο από τις ελληνικές αρχές και από την ελλάδα διευκρινήσεις για μια πρακτική που ακολουθεί το κατά την δεκαετία 1998-2008 από πολλά κράτη μέλη της ευρωζώνης όπως αναφέρεται σε πλήθος δημοσιευμάτων του ξένου τύπου τον τελευταίο καιρό η ελλάδα λοιπόν δεν ζητάει χρήματα ζητάει κάτι άλλο αγαπητές ε, συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφοι κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο όχι μόνο λόγω συμμετοχής στην ευρωζώνη αλλά γενικότερα λόγω συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ένωση την έκφραση μιας πολιτικής υποστήριξης αλληλεγγύης εμπιστοσύνης ουσιαστικής όμως και ειλικρινούς μια υποστήριξη που δεν θα μείνει στα χαρτιά θα έχει ουσία και περιεχόμενο και δεν θα αναιρείται και θα υπονομεύεται μόλις βγαίνουμε από τις κλειστέ αίθουσε. η ελλάδα ζητάει από τους εταίρου να μην δίνουν τροφή με τη στάση και τι δηλώσεις τους στους κερδοσκόπους και να μην σπέρνουν διαρκώ την αμφιβολία για το αν η ελλάδα μπορεί να φέρει αποτέλεσμα με τα μέτρα που εξήγησε. γιατί σε τελευταία ανάλυση με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεται η προσπάθεια που καταβάλει η βόρα. να μην στρουθοκαμιλίζουμε αγαπητέ συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφοι. όλοι γνωρίζουμε ότι οι κερδοσκόποι μέσω της ελλάδας στόχευαν την ευρωζώνη και το ευρώ. ας κινητοποιηθούμε λοιπόν να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για τη θωράκιση της ευρωζώνης και του ευρώ. ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι σήμερα έχουμε μόνο πέντε λεπτά για τη διαδικασία Catch the Eye γιατί μας έχει σωθεί ο χρόνος. Ένα λεπτό αναομιλητή και έχουμε 30 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν έχει νόημα λοιπόν να συνεχίσετε να ζητάτε το λόγο πολύ. Λυπάμαι που σας απογοητεύω. Ο κύριος Δικάστρο, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να εκφράσω τη θλίψη μου και όλη τη Επιτροπή Γεωργία που έχω την τιμή τη Μιζά προεδρεύω γιατί δεν, έλει, δεν αναφέρθηκε καθόλου αγροτικό και τροφιμικό τομέα στη στρατηγική για το 2020. Είναι παράλογο η στρατηγική για τα επόμενα 10 χρόνια που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην συμπεριλαμβάνει το θέμα το κεντρικό τη πρόκληση όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και όσον αφορά την ε, συνάρτηση με την ανάπτυξη τη υπαίθρου και την απασχόληση εκεί. Πώ μπορεί να υπάρχει πράσινη και βιώσιμη Ευρώπη χωρί να λάβουμε υπόψη ότι το 45% όλη τη επικράτεια τη Ευρώπη ε, ε, το χειρίζονται οι γεωργοί. Πώ να μην λάβετε υπόψη σχεδόν 30 εκατομμύρια άτομα που εργάζονται σε αυτή την ε, ύπεθρο. Είναι εργαζόμενοι, πρέπει να προστατεύσουμε πριν ασχοληθούμε με τη νέα απασχόληση, θα πρέπει να υπερασπιστούμε την υφιστάμενη απασχόληση. Υπενθυμίζω ότι η Γεωργία δίνει μια σειρά υπηρεσιών, ουσιοδών, τροφή, βιοπικιλότητα, ύπεθρο, περιβάλλον, ε, λειτουργίε που είναι απαραίτητε για κοινωνική συνοχή, οικονομική συνοχή τη υπαίθρου. Και η Ισπανική Προεδρία επανέλαβε και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει μια κοινή αγροτική πολιτική που είναι ισχυρή. Λοιπόν, ανησυχώ, Πρόεδρε, για αυτή τη σοβαρότατη παράληψη που ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να διορθώσει. Σα ευχαριστώ. Τελευταία ομιλήτρια, η κυρία Γιακονσάρη. Ένα λεπτό έχει επίσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με το κινέζικο ημερολόγιο, έχουμε την χρονιά της τίγρης. Η Ινδία είναι οικονομικός τίγρης και αποτελεί ένα τεράστιο εργοτάξιο. Νομίζω ότι οι εξελίξεις στην Ινδία επηρεάζουν εξαιρετικά και την Ευρώπη. Και χρειαζόμαστε λοιπόν νέα κίνητρα. Χρειαζόμαστε κίνητρα για το 2020. Χρειαζόμαστε μια κοινή οικονομική πολιτική και χρειαζόμαστε επίσης μια τολμηρή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις ε, διαφορετικέ δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Δύο ερωτήσεις έχω να απευθύνω. Τι γίνεται με την ε, ελληνική τραγωδία αυτή, ποια θα είναι τα μαθήματα τα οποία θα εξαγάγουμε για το μέλλον του Συμφώνου Σταθερότητας και κατά δεύτερον τι δυνατότητες έχουμε για την στρατηγική του 2020 προκειμένου να λειτουργήσει καλύτερα για να μην προκληθούν περαιτέρω ελληνικές τραγωδίες. Συνάδελφοι, έχουμε πέντε λεπτά ακριβώς, ε, πέντε ομιλητές και όλοι παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας. Ο κύριος Μαρινέσκου, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, χαίρομαι ιδιαιτέρως που σας βλέπω εδώ στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με καταπλήσευτη η σπουδή του Συμβουλίου να λάβει απόφαση χωρί προηγούμενη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε τη στρατηγική του 2020 γιατί απέτυχε η προηγούμενη στρατηγική τη Λισαβόνα. Τα έγγραφα όμω που κυκλοφορούν είναι πολύ γενικά και αόριστα και, δεν, ε, και μιλούν πολύ γενικά για τι μελλοντικέ προκλήσει. Τι γίνεται με την κοινωνική διάσταση, με τη γύραση του πληθυσμού και την έλλειψη σε ειδικευμένου εργαζόμενου. Λιγότερο από 2% του προπολογισμού αφιερώνεται στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Λάθος κατά τη γνώμη μου και θα πρέπει να διορθωθεί. Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη θα μπορούσαν να στηρίζονται σε συμπράξεις κρατικών και ιδιωτικών κεφαλαίων και να ενθαρρυνθούν οι επιχειρηματίες να επενδύσουν σε εργαστήρια και έρευνα για να αναχαιτήσουμε αυτή τη διαφυγή των εγκεφάλων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνική. Λυπούμε που έφυγε ο πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπής στο μεταξύ, αλλά τουλάχιστον ε, είναι παρόν ο αρμόδιο επίτροπο για τη θεσμική συνεργασία. Για να ευοδοθεί, με ε, να ευοδοθεί η στρατηγική του 2020, για να στεφθεί με επιτυχία, θα πρέπει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να έχουν μια ευγενή άμυλα μεταξύ του και ταυτόχρονα μια αγαστή συνεργασία, προκειμένου να δημιουργηθούν μηχανισμοί για να εφαρμόσουμε τα μέτρα που είναι απαραίτητα. Επίσης θα πρέπει να απαλλαγούμε από τους εθνικούς εγωισμούς και να αναλάβουμε εθνική ευθύνη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλιώς πώς θα μιλούμε για εναρμόνιση της κοινωνικής πολιτικής και της φορολογικής πολιτικής. Αδύνατον να υλοποιήσουμε τους στόχους που σχετίζονται με οικονομική πολιτική προκειμένου να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστική στον κόσμο. Δεν βλέπω να είναι εδώ ο κύριος Στάς, άρα ο κύριος Νταφ παίρνει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων απέναντί σας, διότι περιγράψατε τις προδιαγραφές σας όσον αφορά τη θέση σας. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί αποφεύγεται να απαντήσετε στο κοινοβουλευτικό μου ερώτημα. Σας παρακαλώ να το επανεξετάσετε το θέμα, να επανεξετάσετε την προσέγγισή σας όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και ζητώ συγγνώμη για την τροπιαστική συμπεριφορά του Νάιτζολ Φάρατζ. Και σας εγγυώμαι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Βρετανών Ευρωβουλευτών θα σας αντιμετωπίσουν με κάθε σεβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε το τελευταίο διάστημα τα μάτια όλη τη Ευρώπη και όχι μόνο είναι στραμμένα στην ελλάδα και το είπαν προηγουμένω και πολλοί ομιλητέ. σε ένα περιβάλλον παγκόσμια οικονομική κρίση, βεβαίω, δεν είναι μόνο η ελλάδα που έχει σοβαρό πρόβλημα οικονομικό είναι και άλλε χώρε και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. είμαστε μάρτυρε μια πρωτόγνωρης κερδοσκοπική επίθεση που εσχάτω και λυπάμαι γι' αυτό πήρε τη μορφή συκοφαντία και μάλιστα του χειρίστου είδου από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωση σε κάθε περίπτωση και να είστε όλοι σίγουροι γι' αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η ελλάδα δεν χρεοκοπεί η ελλάδα δεν καταραίει. άλλωστε ποτέ η χώρα μας δεν ζήτησε οικονομική βοήθεια. αυτό που ζήτησε και ζητάει είναι πολιτική στήριξη. αυτό που ζήτησε και ζητάει είναι η έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης των υπολείπων κρατών μελών στα πλαίσια της ε, ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης την οποία και έχουμε γιατί τελικά αυτό είναι το διακύβευμα. σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις αρχές του έτους ε, η ανεργία ανέβηκε για παραπάνω από 10% και το ανέβηκαν επίσης, αυξήθηκαν και τα δημοσιονομικά χρέη. Οι Ευρωπαίοι πολίτε ζητούν απαντήσει σε όλα τα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύσει κατά προτεραιότητα στη δημιουργία θέσεων εργασία στην ανάπτυξη υποδομών, στην εκπαίδευση, στην γεωργία. Χρειάζεται επίσης μία βιώσιμη στρατηγική για την ενέργεια και θα πρέπει να επενδύσουμε στην ενεργειακή αποδοτικότητα σε ό,τι αφορά τις κατοικίες αλλά και σε ό,τι αφορά τις βιομηχανίες. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2020. Επίσης θα πρέπει να επενδύσουμε στις βιομηχανίες εντός της Ένωσης, όχι μόνο να επιτρέψουμε και να αφήσουμε την μετεκατάσταση των επιχειρήσεων. Επίσης θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν τα κοινωνικά συστήματα για να εγγυούμαστε την ε, αξιοπρεπή διαβίωση όλων των πολιτών. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, κλείνουμε τώρα τη συζήτηση. Πρώτα με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον ε, του κ. Σεύκοβιτς. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σημερινή σύνοδο ξεπέρασε τα χρονικά όρια και ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να αποχωρήσει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Αν είναι τιμή για μένα πραγματικά να απαντήσω εκ μέρου του Προέδρου Μπαρόσο και εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα όλου σα για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, με πολύ ενδιαφέρουσε ιδέε και με μεγάλο ενθουσιασμό και υποστήριξη που δείξατε προς την ε, στρατηγική για το 2006 Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χωρίς την υποστήριξή σας δεν θα πετύχει αυτή η στρατηγική για το 2020. Σας διαβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πολύ τολμηρή θα βάλουμε τον πολίτη, την απασχόληση, τη μείωση της φτώχειας ε, στο επίκεντρο της πολιτικής για το 2020. Σας διαβεβαιώνω ότι μάθαμε τα μαθήματά μας από τη στρατηγική της Λισαβόνας και γι' αυτό θα εστιαστούμε επί μικρότερου αριθμού στόχων και σίγουρα θα βελτιώσουμε τη διαχείριση τη στρατηγική και τη διακυβέρνηση. Ενθαρρύνεται πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μεγάλο ενδιαφέρον και ελπίζουμε μεγάλη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενθαρρυνόμεθα τα μάλα και από τι είδαμε ότι στο Συμβούλιο θέλουν να κινηθούμε γρήγορα, αλλά η σημερινή ατμόσφαιρα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι πριν από μια πενταετία όταν συζητούσαμε τι παραμέτρου στρατηγική τη Όμω, θα κάνουν περισσότερα. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των λαών για τη στρατηγική. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες θα το δουν σαν ένα διοικητικό εγχείρημα, αλλά μια προσέγγιση που θα βελτιώσει τη ζωή στην Ευρώπη και στις χώρες τους και στις περιφέρειές τους. Και θα ήθελα να σας ζητήσω αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας βοηθήσετε για να εκτελέσουμε αυτό το καθήκον. Α μην υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων, αλλά συνεργασία. Συστιαστούμε επί των προτεραιοτήτων και πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στη στρατηγική για το 2020 Ευρωπαϊκή Ενώσεω θέλουμε να εισαγάγουμε τρει πυλώνε. ΕΦΗ, πράσινη, ενταξιακή οικονομία θέλουμε. Και θέλουμε να βασιστούμε στου τρει πυλώνε. Θα πρέπει να δρομολογήσουμε πρωτοβουλίες που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας που μπλοκάρουν την οικονομία και δεν μπορεί να αναπτυχθεί στο πλήρε δυναμικό τη. Θα πρέπει να στεστούμε επιπαιδείας καταρτήσεω, ώστε το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη να είναι ανταγωνιστικότερο έναντι των άλλων. Αυτό το αξίζει η Ευρώπη. Η στρατηγική για το 2020 της Ευρώπης θα συνδέεται με το Σύμφωνο για Σταθερότητα και την Ανάπτυξη. Χρειάζεται μια στεναρή φορολογική πολιτική. Είναι βασικό στοιχείο για τη σταθερότητα της οικονομίας. Ε, μιλήσαμε πολύ για την Ελλάδα σήμερα και σας διαβεβαιώνω ότι υπήρξε συνένεση ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα πάρουν αποφασιστικά και συντονισμένα μέτρα και δράση αν αυτό χρειαστεί για να διαφυλάξουν την οικονομική σταθερότητα στον τομέα της Ευρωζώνης στην Ευρωζώνη και θα συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ελλάδα και θα παρακολουθήσει πώς εφαρμόζει η Ελλάδα τις συστάσεις. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Εθνές Νομισματικό Ταμείο συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Υπάρχει αποστολή των τριών φορέων στην Αθήνα που θα βοηθήσει την Ελλάδα να πάρει συμπληρωματικά μέτρα. Έχουμε τα εργαλεία για να προφυλάξουμε την οικονομική σταθερότητα τη Ευρωζώνη αν αυτό χρειαστεί. Αυτό συνεπάγεται ότι θα συνεργαστούν τα μέλη τη Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το συντονισμό των δράσεων σε κάθε στάδιο. Όμω θα πρέπει να δώσουμε τον κατάλληλο χρόνο. Εξαρτάται τώρα από την Ελλάδα να κάνει η Ελλάδα τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να πάρει τα αναγκαία μέτρα. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα τολμηρά βήματα ε, και όσον αφορά τη θετική το 2020 και όσον αφορά την κατάσταση που στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κύριος ε, Βανόμπαϊ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερως για τη δυνατότητα που είχα να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση και χαίρομαι που δέχτηκα την πρόσκλησή σας να έρθω εδώ στην αρχή της διαδικασίας αυτής για τη στρατηγική του 2020. Γιατί μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στα σπάργανα της συζήτησης, στην απαρχή της διαδικασίας. Έγινε μια συζήτηση στις 11 Φεβρουαρίου. Ακολουθεί το Εαρινό Συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου και θα οριστικοποιηθεί η στρατηγική του 2020 για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη τον Ιούνιο. Έχουμε μία μακρά περίοδο για ανταλλαγή απόψεων και για την ε, για τον ακριβή προσδιορισμό των δράσεών μας. Χαίρομαι για την ευρωπαϊκή φιλοδοξία που διέγνωσε σήμερα το απόγευμα από τη συζήτηση και χαίρομαι για τις φιλοδοξίες σας και για την αίσθηση που έχετε ότι η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Και για μία παρέμβαση μόνο περιφρόνηση μπορώ να εκφράσω, απαξιό όμως δεν πρόκειται να επανέλθω σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά την οικονομική στρατηγική έκανα μια διάκριση μεταξύ τριών περιόδων. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη φάση, είναι η φάση που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τη χρηματοπιστωτική κρίση με τις συνέπειές της. Και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια άλλη ορολογία από αυτή που άκουσα το απόγευμα καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μια θετική διατύπωση. Γιατί υπάρχουν και θετικά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θετικές εξελίξεις τον τελευταίο καιρό. Αντλήσαμε κάποια διδάγματα και διδαχθήκαμε από τα παθήματα της κρίσης του 30. Έχει περάσει ένας χρόνος μετά τη μεγάλη κρίση. Και σήμερα, το 2010, στις περισσότερες χώρες διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Κάτι που δεν συνέβη στη δεκαετία του 30. Εκεί η κρίση κράτησε μια ολόκληρη δεκαετία. Γιατί λοιπόν έχουμε τώρα θετική ανάπτυξη. Έχουμε θετική ανάπτυξη γιατί λάβαμε κάποια μέτρα. Μέτρα για να σώσουμε τα χρηματοπιστωτικά όργανα. Όχι γιατί τα υπεραγαπούμε, αλλά χωρίς ε, χρηματοπιστωτικά όργανα, χωρίς τράπεζες ε, δεν υπάρχει τέτοια οικονομική πολιτική. Ταχθήκαμε υπέρ μια ευφυού νομισματική πολιτική. Βελτιώσαμε τη ρευστότητα, κάτι που δεν έγινε πριν από 70 χρόνια. Για 16 τουλάχιστον χώρε δημιουργήσαμε μια ζώνη, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, μια ζώνη νομισματική σταθερότητα. Στη δεκαετία του 30 είχαμε ανταγωνιστικέ υποτιμήσει, κάτι που δεν συνέβη σήμερα εφαρμόσαμε μία αρκετά παρακινδυνευμένη δημοσιονομική πολιτική, χρησιμοποιώντα τα δημοσιονομικά ελλείμματα για να δώσουμε ενάψματα στην οικονομία. Κάτι που δεν συνέβη στη δεκαετία του 30, που προσπαθήσαμε το συντομότερο δυνατό να επανέλθουμε σε μία δημοσιονομική ισορροπία. Διαφυλάξαμε, διαφυλάξαμε, επαναλαμβάνω, την εσωτερική μας αγορά, που δεν είναι τέλεια και χρήζει εμβάθυνση. Γι' αυτό και ο Επίτροπο Μόντι θα υποβάλει, ο κ. Μόντι θα υποβάλει συγκεκριμένε προτάσεις. Αλλά δεν ενδώσαμε στον προστατευτισμό της δεκαετία του 30. Οπότε διδαχθήκαμε από τα παθήματα της μεγάλη κρίση που βιώσαμε. Και θα έλεγα και κάτι παραπάνω. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε το G20. Εμείς αναλάβαμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε αυτό το φυτόριο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Για πρώτη φορά οι υπερδυνάμεις, οι παλιές και οι καινούργιες, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι για να καταπολεμήσουν την κρίση. Ναι, με ατελή τρόπο, αλλά θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στην άμυνα. Δεν θα πρέπει να παίζει πάντα αμυντικό παιχνίδι. Γιατί υπάρχουν και πολύ γεγονότα και πολύ θετικές εξέλιξεις. Τώρα, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια στρατηγική εξόδου από την κρίση και να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ του να καταλήψουμε πολύ γρήγορα τα δημοσιονομικά ενάυσματα και ταυτόχρονα μέσω πρόθεσμα να επανέλθουμε σε μια δημοσιονομική ισορροπία που είναι απολύτως απαραίτητη για να, για να χρηματοδοτήσουμε τα συνταξιοδοτικά μας συστήματα και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και υγειονομικής περίθαλψης. Θα πρέπει να βρούμε αυτή την ε, λεπτή και εύθραυστη ισορροπία. Και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μας δίνει τα μέσα για κάτι τέτοιο, γιατί δεν ζητά άμεση επιστροφή στην δημοσιονομική ισορροπία, αλλά ζητά προοδευτικά, βήμα με βήμα, να φτάσουμε πρώτα στο 3% και μεσοπρόθεσμα να υλοποιήσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία. Νομίζω ότι θα προλάβουμε και θα έχουμε το χρόνο να υιοθετήσουμε μια συνετή και φρόνιμη πολιτική. Σε ό,τι αφορά τώρα τη στρατηγική της Λισαβόνας. Γνωρίζουμε τις αδυναμίες της στρατηγικής της Λισαβόνας. Αλλά α μην ξεχνούμε ότι η χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική κρίση διατάραξαν τα μάλα την ε, υλοποίηση του προγράμματος της Λισαβόνας. Αλλά υπήρχαν κάποια κενά, κάποιες αδυναμίες γνωστά σε όλους δεν πρόκειται να τα απαριθμίσουμε τώρα όλα αυτά. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι χρειάζονται ρηξικέλευθε μεταρρυθμίσεις, ή τουλάχιστον πολύ σημαντικέ μεταρρυθμίσεις. Και αυτέ οι σημαντικέ μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν και σε πανευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Κάτι που προποθέτει κάποιε δημοσιονομικέ επιλογέ. Δεν είναι τυχαίο που στα συμπεράσματα που σα έστειλα στην επιστολή μου, δεν είναι τυχαίο που συνδέουμε την δημοσιονομική συζήτηση στο νομικό πλαίσιο φυσικά του Συμφώνου σταθερότητα με τι οικονομικέ μεταρρυθμίσει. Γιατί αν πούμε ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, θα πρέπει να το προβλέψουμε και στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στις δημοσιονομικές προοπτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει συγκεκριμένες δημοσιονομικές επιλογές. Μία άλλη επίπτωση των επιλογών μας για τη στρατηγική της Λισαβόνας όλοι οι στόχοι που προτείνουμε δεν είναι πάντα ήπιοι στόχοι. Μπορεί να είναι και σκληροί στόχοι. Και εκεί θα έρθουν τα ζόρια. Γιατί υπάρχει απέτηση μεταρρυθμίσεων, αλλά υπάρχει και η φάση της εκτέλεσης των μεταρρυθμίσεων, της εφαρμογής τους. Δεν το άκουσα και πολύ εδώ. Γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτός του Κοινοβουλίου, απαιτούνται αυστηρά μέτρα, σκληρά μέτρα, δρακόντια μέτρα και μεταρρυθμίσεις, αλλά όταν επιστρέφει κάποιο στη χώρα του βλέπω ότι ελάχιστα είναι τα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε όμως συνέπεια μεταξύ αυτών που ζητούμε και αυτών που κάνουμε. Δεν πρόκειται μόνη της Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει όλες τις μεταρρυθμίσεις. Μπορεί να εμψυχώσει τα κρατημέλη, να τα ενθαρρύνει, να τα παροτρύνει, να πλαισιώσει τις μεταρρυθμίσεις, αλλά οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο. Και κάτι τέτοιο προϋποθέτει μία δεδηλωμένη πολιτική βούληση. Και η πολιτική δέσμευση είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Πολύ συχνά λέμε ότι χρειάζονται πιο δεσμευτικά μέτρα. Ας το σκεφτούμε όμως. Έχω υποβάλει πολλοί άριθμες πρότασεις και νομίζω ότι είναι πιο έξυπνες από κάποια δεσμευτικά μέτρα ακόμη και το σύμφωνο σταθερότητας, που περιλαμβάνει και δεσμευτικά μέτρα, δεν κατόρθωσε να επαναφέρει στην τάξη ορισμένες χώρες. Οπότε δεν αρκεί η μέθοδος. Η μέθοδος δεν είναι πανάκια. Η μέθοδος χωρίς πολιτική δέσμευση είναι κενό γράμμα. Για την οικονομική στρατηγική, μερικοί μου λένε χρειάζεται πιο μεγαλύτερη δέσμευση, υποχρεωτικό χαρακτήρα, Αλλά για τις οικονομικές κατευθυντήρε γραμμέ, η συνθήκη τη Λισαβόνα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Δεν είναι δική, δικό μου δημιούργημα η συνθήκη τη Λισαβόνα. Άλλοι το, την έφτιαξαν και δεν προβλέπονται ούτε κυρώσεις, ούτε ε, αρνητικά μέτρα για την εφαρμογή των ε, οικονομικών κατευθυντήριων γραμμών και σας παραπέμπω στο άρθρο 121 για να βεβαιωθείτε για αυτό που σας λέω. Χρειάζεται πολιτική δέσμευση και ανάληψη ευθύνης και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χωρίς τέτοια πολιτική δέσμευση τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Και τέλος για την Ελλάδα. Δύο λόγια. Νομίζω ότι ήταν σωστό το μήνυμα που διαβιβάσαμε. Νομίζω ότι πέρασε το μήνυμα της ευθύνης της ελληνικής κυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να χειριστεί μια εξαιρετικά χαλεπή κατάσταση. Μια κατάσταση που έχει εκνευρίσει. Θα κληθεί η ελληνική κυβέρνηση να λάβει πολύ θαραλέα και τολμηρά μέτρα. Στις 11 Φεβρουαρίου μας είπαν ότι αν δεν αρκέσουν αυτά τα μέτρα για να μειωθεί κατά 4% το δημοσιονομικό έλλειμμα στο ΕΠ, το 2010 θα λάβουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Και δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για περισσότερη παρακολούθηση και εποπτεία. Όχι μόνο με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και με ε, πυρογνωμοσύνη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεσμεύτηκε για περισσότερη εποπτεία. Νομίζω ότι πλαισιώσαμε και περιορίσαμε με πολύ σωστού όρου το θέμα της ευθύνη. Φυσικά, αν χρειαστεί, υπάρχει και το στοιχείο της αλληλεγγύη. Η Ελλάδα μας είπε ότι δεν θέλω να απευθύνω έκκληση στην αλληλεγγύη σα. αλλά προβλέψαμε δύο μήνυματα. Το μήνυμα της ευθύνης, αλλά και το μήνυμα της αλληλεγγύη, αν παραστεί ανάγκη. Και φυσικά θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα από όσα συνέβησαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και στην Ευρωζώνη θα πρέπει να είμαστε πιο δραστήριοι και στην συλλογή των δεδομένων αλλά και στην άσκηση της πολιτικής. Αυτή η κρίση όμως ήταν μια πρόκληση για όλους μας. Μια πρόκληση που μας έδειξε ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε περισσότερο την πολιτική συντονισμού. Κάθε κρίση δημιουργεί και μια πρόκληση και κάθε κρίση θα πρέπει να μας διδάσκει ορισμένα πράγματα. Όπως αντιλήσαμε διδάγματα από την κρίση της δεκαετίας του 30, θα εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα και από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ρύθμιση, περισσότερο έλεγχο των πόνους, περισσότερη ε, τραπεζική πολιτική. Και φυσικά θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα και από την ελληνική εμπειρία και άλλες εμπειρίες. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αισθάνθηκα εδώ την ίδια φιλοδοξία και την ίδια πολιτική βούληση για την εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής και οικονομικής στρατηγικής που θα σταθεί στο ύψος των δυσκολιών μας και θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Και αυτό δεν είναι ευθύνη ενός ή δύο ανθρώπων. Θα πρέπει να αναλάβουμε συλλογικά αυτή την ευθύνη. Όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει από κοινού να αναλάβουν την ευθύνη. Αλλιώς δεν θα διαφυλάξουμε το κοινωνικό μας μοντέλο θα χάσουμε τη θέση μας στον κόσμο. Και με αυτό το πνεύμα ήρθα σήμερα το απόγευμα να σας μιλήσω και με, με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσω και το έργο μου. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν μεγάλη τιμή που παρευρεθήκατε εδώ στη συνεδρίασή μας, ε, στην παρθενική σας εμφάνιση εδώ στην Ολομέλεια, στην ε, Ελλάδα. Έχουμε ε, την έκφραση συντροκέφαλος σιδερό κεφάλι σας εύχομαι λοιπόν για να αντέξετε όλα όσα θα επέλθουν σε μια δύσκολη πορεία. Νομίζω ότι καταδείξατε ότι μπορείτε να το κάνετε αυτό και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που βρεθήκατε εδώ σήμερα. Η μερίσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου εν ώψη της Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Γενέβη, 1 με 26 Μαρτίου 2010. Αρχίζουμε τη συζήτηση εξ του Συμβουλίου. Θα δώσουμε ένα λεπτό περίπου.